Ο Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε. Ε, Δεν έχω ανακοινώσει να κάνω ε, επί της ημερησίας διατάξεως. Άρα το τρίτο θέμα είναι η παρουσίαση του σύντομου ενημερωτικού σημειώματος για την αξιολόγηση των αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου στην Ευρώπη, την οποία θα μας κάνει η κόβη, καλωσορίζω τους ε, κυρίους Χάντζεν και Πέτερσεν. Έχουμε προβλέψει μία ώρα για την συζήτηση αυτή. Πώς λέτε να αρχίσετε. Κυρία Χάνσεν. μπορείτε να αρχίσετε. Σας ευχαριστώ. Λέγομαι Τίνα Χάνσιν από την Δανική Κόβη. Έχουμε έδρα τη Δανία και παρέχουμε συμβουλές για θέματα περιβαλλοντικά. Σύντομη εισαγωγή. Το σημείωμά μας μας ζητήθηκε να είναι σύντομο και περιεκτικό, να δώσει ιδιαίτερο βάρος στα τεχνικά και πολιτικά θέματα που έχουν σχέση με τους αγωγούς αερίου και πετρελαίου βασιζόμενο στα υφιστάμενα έγγραφα και στην ε, ε, υφιστάμενη ε, βιβλιογραφία. Άρα υποτίθεται ότι ανταποκρίνεται, είναι επίκαιρο το, το σημείωμα μας αυτό. Επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο στον συναδελφό μου κύριο Πέτερσεν, που είναι οικονομολόγος ενέργειας στην COVID για να περάσει τις λεπτομέρειες της παρουσίασης. Σας ευχαριστώ. Η παρουσίαση ακολουθεί ακριβώς και το σημείωμα. Συζητούμε δηλαδή τις αλυσίδες παροχής, μπαίνουμε ε, λίγο ε, στην υποδομή και συζητούμε ορισμένα επιμέρους θέματα και μετά προβλέπουμε χρόνο για ερωτήσεις και απαντήσεις. εξετάζουμε την υποδομή, δεν συζητούμε την μαλακή πλευρά, δηλαδή το ίδιο το αέριο, μόνο την υποδομή. Υπάρχουν κάποιοι, κάποιες διαφορές ανάμεσα σε πετρελαγωγούς και αγωγούς φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο συνήθως, ε, ο αγώστος δηλαδή, συνδέεται με την πηγή και συνήθως καταλήγει στην παγκόσμια αγορά ή στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου καθορίζει τη τιμή του φυσικού αερίου. Το αέριο είναι ανελαστικό στην ζήτηση και στους αγωγούς. Μπορεί να παράγεται LNG ή CNG που είναι κάπως πιο ελαστικό. Για, τον, για την αγορά πετρελαίου τα πράγματα είναι πιο απλά. Η μεταφορά και η αποθήκευση είναι και πιο ελαστικές και πιο εύκαμπτες δηλαδή, αλλά και πιο εύκολες και είναι και πολύ διαφορετικές οι μέθοδοι μεταφοράς και αποθήκευσης ε, ανάμεσα στα δύο αυτά είδη ενέργειας και γι' αυτό και ο ανταγωνισμός είναι και μεγαλύτερος και στην περίπτωση του πετρελαίου εφαρμόζονται οι ε, κανόνες ανταγωνισμού της Ένωσης και αυτό ισχύει και για την υποδομή ενώ για το η πρόσβαση στην υποδομή του αερίου είναι κανονιστικά ρυθμισμένη. Βλέπετε το χάρτη των υφισταμένων και υποσχεδιασμό αγωγών και των υπολείπων τμήματων της υποδομής Επί του παρόντος το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται κατά 500 εκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου τον χρόνο και πρόκειται να αυξηθεί με τον χρόνο αυτό, το έτος δηλαδή, πρόκειται να αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου, αν και και τα πιο αισιόδοξα σενάρια για την χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας δείχνουν ότι και σε 20 χρόνια το καταναλούμενο αέριο θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα. Η παραγωγή αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να μειωθεί από 200 σε 100 περίπου δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Με την αυξανόμενη ζήτηση και με τις περισσότερες αγωγές θα χρειαστούν, με την δηλαδή, θα χρειαστούν και αυξήσεις στις επενδύσεις της υποδομής η ικανότητα εισαγωγής είναι επαρκής για την ώρα υπό κανονικές συνθήκες. Αλλά με την αναμενόμενη αύξηση θα χρειαστεί να γίνουν και νέες επενδύσεις σε υποδομές. Το κενό μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης σήμερα καλύπτεται κυρίως από τις εισαγωγές από τη Ρωσία, την Νορβηγία και από τη Συρία, αλλά και από υγροποιημένο αέριο και από την Νορβηγία. νέα project εισαγωγής και διασύνδεσης θα χρειαστούν στο μέλλον για να, αυξηθεί, να αυξηθούν οι ικανότητες εισαγωγής. Έχουμε σήμερα και το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Έχουμε σχετικές εγκαταστάσεις και είναι και μια δυνατότητα αυτή διαφοροποίησης μέσα στο σύστημα. Πιο μακροπρόθεσμα η εστίαση θα μετατοπιστεί προς αποθέματα που ίσως είναι πιο, θέματα που είναι πιο μακριά, όπως στη Ρωσία, στο Ιράν, στο Κατάρ και στη Μέση Ανατολή. Έχουμε για την ώρα τρεις ή τέσσερις περιοχές για το αέριο στην Ευρώπη. Έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή έχουμε τη Βόρεια, περιοχή, τη νότιο-ανατολική και την νότιο-δυτική. Και σε ορισμένες περιπτώσεις και η Βαλτική και η Φιλανδία θεωρούνται μια ξεχωριστή περιφέρεια. Τα κριτήρια για, την, για τις περιφέρειες αυτές είναι και η προέλευση της πηγής, αλλά και η γεωγραφική απόσταση και οι δυνατότητες ε, να γίνει pooling στις ε, εγκαταστάσεις αποθήκευσης του αερίου. Ο πιο σημαντικός διάδρομος είναι ο βορειοανατολικός από τη Ρωσία με 23% της κατανάλωσης, δηλαδή που παρέχει 24% της κατανάλωσης. Υπάρχει και ο βορειο διάδρομος από την Ορβηγία και καλύπτει 18 περίπου της 100. Ο νοτιο από την Αλγερία περίπου 10%. και ενδεχομένως και ένα διάδρομο νότιο-ανατολικό που πιο μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να αποτελέσει μια νέα δίωδο προμήθειας μέσα στα πλαίσια μιας προσπάθειας διαφοροποίησης το εσωτερικό δίκτυο μεταφοράς είναι ιδιαίτερα πυκνό στην, στις βόρειες περιφέρειες Ολλανδία, Βέλγιο όπου έχουμε υψηλή πυκνότητα ε, αγωγών μεταφοράς δυνατότητες υπόγειας αποθήκευσης Εκεί τέτοιες έχουμε κυρίως στη Γερμανία, Ιταλία και Αυστρία με υψηλή δυνατότητα αποθήκευσης. Λείπουν όμως τις περισσότερες από τις άλλες χώρες. Το σύστημα είναι σχετικά νέο σε ηλικία και λειτουργεί καλά. Υπάρχει και ένας αριθμός νέων αγωγών που πρόκειται να κατασκευαστούν ένας από τον Νότο, Green Stream μεταξύ δηλαδή Λιβύης και Ιταλίας περνώντας από Σικελία, νέους αγωγούς μεταξύ ενδεχομένως Ολλανδίας και ε, Ηνωμένου Βασιλείου, άλλον αγωγό μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος και υπάρχουν υποσχεδιασμό ορισμένα έργα από Αλγερία την Ισία Σικελία Ιταλία, από Αλγερία Ισπανία, μεταξύ Ρωσίας-Γερμανίας επίσης και μεταξύ Αλγερίας-Ιταλίας μέσω Σαρδινίας αυτή τη φορά. Και έχουμε και τον αγωγό Ναμπούκο που υποτίθεται ότι θα συνδέσει την Κασπία στην Κεντρική Ασία με την Μέση Ανατολή μέσω Τουρκίας. Αυτά τα νέα σύστημα, συστήματα συγγνώμη, αγωγών θα αυξήσουν κατά 90 περίπου ε, δισεκατομμύρια κυβικών μέτρων τα επόμενα χρόνια της δυνατότητες μεταφοράς αερίου. Εν συνόψη το βασικό πρόβλημα εν προκειμένου είναι ότι υπάρχει το κενό αυτό μεταξύ κατανάλωσης και παραγωγής που χρειάζεται κατασκευή νέων ε, αγωγών, νέα σχήματα παροχής όπως λέχθηκε και πριν, ενίσχυση των υφιστάμενων διαδρόμων μεταφοράς και βεβαίως νέες υποδομές. Η πολιτική, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020, 20, για τη μείωση δηλαδή των διοξιδίων ε, του ανθράκος, θα επηρεάσει την κατανάλωση του αερίου, θα αυξηθεί η ζήτηση, γιατί θα χρησιμοποιηθούν περισσότερα εργοστάσια που καίνε αέριο για να ε, γίνει σταδιακή κατάργηση των, ε, του άνθρακα, της χρήσης του άνθρακα δηλαδή, αλλά είναι ακόμα ανοιχτό, μένει ακόμα ανοιχτό το ερώτημα πώς δηλαδή οι προσπάθειες καταπολέμησης των αρνητικών επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος θα επηρεάσουν την ε, ζήτηση του αερίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους πετρελαιαγωγούς, έχουμε εισαγωγές μέσω αγωγών. Έχουμε και έναν από τους μακρότερους πετρελαγωγούς του κόσμου που έρχεται από τη Ρωσία και προμηθεύει μέσω τριών κλάδων προς βορρά, προς το κέντρο και προς νότον το ανατολικό μέρος της Ευρώπης. Πάει στη Λευκορωσία, την Πολωνία. και στην Σλοβακία. Ο άλλος σημαντικός αγωγός έρχεται από την Νορβηγία η, του πρώτου η ικανότητα μεταφοράς είναι 100 εκατομμύρια τόνων τον χρόνο. Δεν εξαντλείται. Βρίσκεται σε περίπου στα 65 αυτή τη στιγμή. 65 εκατομμύρια τόνους τον χρόνο. Για το λόγο αυτό η Ρωσία σχεδιάζει να μεταφέρει κάποιες από τις προμήθειες αυτές και στην Ανατολική Ευρώπη Κάτι που ίσως να οδηγήσει σε κάποιες συνέπειες στην προμήθεια εκεί. Άλλος σημαντικός αγωγός είναι ο βόρειος από, από την Νορβηγία στο T-side του Ηνωμένου Βασιλείου. Περίπου 4 εκατομμυρίων τόνων ικανότητας μεταφοράς. Μέσα στην Ένωση τώρα, εδώ βλέπετε έναν χάρτη των διαφόρων πετρελαγωγών, με μήκος 33.000 χιλιόμετρων το πιο σημαντικό στοιχείο για το μέλλον είναι ότι υπάρχει μια μικρή διασύνδεση μόνο στο κέντρο της Ευρώπης, κοντά στην Ingolstadt δηλαδή, που συνδέει τα δύο συστήματα. Είναι δηλαδή στην ουσία τα δύο συστήματα χωριστά. Με τα δύο συστήματα πετρελαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η περιορισμένη δηλαδή διασύνδεση είναι ένα σημαντικό στοιχείο για το μέλλον ανάμεσα στους δύο αγωγούς, τον Ανατολικό και τον Δυτικό. Και για την ασφάλεια των προμηθειών, κυρίως του ανατολικού μέρους της Ευρώπης, παίζει σημαντικό ρόλο. Και η ρωσική πολιτική ασφαλώς επηρεάζει σημαντικά το ανατολικό μέρος. Υπάρχουν υποσχεδιασμό και ορισμένα νέα έργα κατασκευής πετρελαγωγών, ένα από την Κωνσταντσα στην Τριέστη, από το Μπουργκάς στο Βλόρε, και στην Τουρκία υπάρχει ένα άλλο και από την Οδυσσό στο πολωνικό Γκτάνσκ. Τα έργα αυτά θα επιτρέψουν μια διαφοροποίηση των διαδρομών του πετρελαίου. Ο 80% ένα μικρό μέρο, ένα μικρό μέρο μόνο των προϊόντων πετρελαίου περνά από του αγωγού και ότι 80% ε, ε, μεταφέρονται με οχήματα, με σκάφη, με πλοία δηλαδή και με σιδηροδρόμους. Είναι αδύναμη διασύνδεση μεταξύ των δύο συστημάτων Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης. Η Ανατολική Ευρώπη είναι τρωτή απέναντι στις ε, προσπάθειες της Ρωσίας να χρησιμοποιήσει τις προμηθείες πετρελαίου για άλλους στόχους το πετρέλαιο θα έπρεπε να περιληφθεί στην ε, εσωτερική αγορά για λόγους ασφάλειας των ε, προμηθειών. Είπα πριν ότι η αγωγή αερίου είναι πιο περίπλοκη υπόθεση. Τα συστήματα αερίου χρειάζονται και μεγάλες αποθήκες για να μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά περισσότερο από ότι το πετρέλαιο δηλαδή, υπάρχουν περιορισμοί και εσωτερικά στην Ένωση, κυρίως για την ροή αποθηκεύσεων και αυτό επηρεάζει την ασφάλεια προμηθειών σε ορισμένες χώρες, για παράδειγμα μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας, αλλά και στην κεντρική Ευρώπη, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία, Αυστρία και έχουν και τη δυνατότητα αντιστροφής της ροής οι τεχνικές προδιαγραφές και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στις διάφορες χώρες μέλη διαφέρουν και αυτό επηρεάζει πάλι τις ε, καθημερινές λειτουργίες. Εξαρτάται πώς εξισορροπούν τη λειτουργία των συστημάτων οι χώρες μέλη. Μιλούμε πάντα για το αέριο. Και πώς χρησιμοποιούνται οι ικανότητες αποθήκευσης. Όλα αυτά βέβαια έχουν επιπτώσεις στην ολοκλήρωση της αγοράς αυτής. Από την οικονομική σκοπιά οι αγωγοί έχουν το, παρουσιάζουν το πρόβλημα ότι είναι σταθερά εγκυρωμένοι ανάμεσα σε δύο σημεία, δεν έχουν εναλλακτικές χρήσεις, είναι υψηλό το κόστος ε, της αρχικής επένδυσης και χαμηλό το κόστος λειτουργίας η αγορά για μεταφορές πετρελαίου θεωρείται ανοιχτή, ενώ του αερίου είναι κανονιστικά ρυθμισμένη. Για την μεταφορά του αερίου δηλαδή. Και η πρόσβαση από τρίτα μέρη ε, και οι σχετικοί κανόνες εφαρμόζονται σε ολόκληρο το σύστημα των αγωγών αερίου. Για να αυξηθεί η ασφάλεια προμήθειας και για να αναπτυχθεί η αγορά του φυσικού αερίου πρέπει να βελτιωθούν τα δίκτυα, να είναι πιο αποτελεσματικές οι διαδικασίες, οι υπερεθνικές διαδικασίες ε, κατανομής των παροχών. Υπάρχουν και ανησυχίες σχετικές με την ασφάλεια των μεταφορών που έχουν σχέση με τις ε, διαδρομές που καλύπτουν οι αγωγοί όταν περνούν από χώρες όπου σημειώνεται αστάθεια και υπάρχει και το ερώτημα που σας είπα και πριν. Οι εσωτερικές διασυνδέσεις και τα σημεία όπου σημειώνονται οι διασυνδέσεις παίζουν σημαντικό ρόλο για την ασφάλεια των προμηθειών, αλλά και για τον μελλοντικό ανταγωνισμό μέσα στην αγορά αερίου. Βλέπετε στο χάρτη τα υφιστάμενα και τα μελλοντικά σημεία εισαγωγής για το φυσικό αέριο. Τα υφιστάμενα είναι τα ακιανού χρώματος. Έχουμε τα, σε μαύρο χρώμα τα υφιστάμενα και σε κόκκινο τα μελλοντικά. και βλέπετε στο χάρτη αυτό ότι ιδίω στο ανατολικό μέρος της Ένωσης υπάρχει ανάγκη να αυξηθούν τα σημεία διασυνδέσεως και με αντιστροφή της ροής και με διαφοροποίηση, αλλά και σε χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Γαλλία πάλι. Υπάρχει και εκεί δηλαδή η ανάγκη να ενισχυθεί η υποδομή. Οι νέες ε, διασυνδέσεις γίνονται λόγω των αναγκών ασφάλειας ε, των προμηθειών, της ανάπτυξης της αγοράς και βέβαια το ερώτημα είναι ποιος θα αναλάβει τις επενδύσεις αυτές που δεν είναι όλες βιώσιμες και κυρίως στο ανατολικό μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ίσως υπάρχει ένα πρόβλημα με την εμπορική βιωσιμότητα των νέων αυτών σημείων διασύνδεσης. υπάρχει και ανάγκη εναρμόνισης των προδιαγραφών. Και η διαφοροποίηση των πηγών είναι σημαντική. Και πρέπει να αρχίσουν να εφαρμόζονται, πρέπει να αρχίσουν να υλοποιούνται τα μεγάλα αυτά έργα υποδομών όπως ο αγωγός Ναμπούκο σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ε, συμβάλλουν και οι εξαγωγείς. Τέλος έχουμε εξετάσει τις διασυνδέσεις και με απομονωμένες περιφέρειες. Υπάρχουν δύο απομονωμένες περιφέρειες. που σημειώνουμε στο σημείωμα μας είναι οι Βαλτικές χώρες και η Φιλανδία και το βόρειο μέρος της, ε, Πολανδία, ε, της Πολωνίας και η κεντρική Σουηδία και πολλά από τα νησιά στην Ένωση θεωρούνται απομονωμένες περιφέρειες σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της χρήσης του αερίου και χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή εκεί θα προκύψουν και πολλά πλεονεκτήματα και για την απασχόληση αλλά και για την ε, βιομηχανική ανάπτυξη και για την προστασία του περιβάλλοντος εφόσον καταστεί δυνατό να ενισχυθεί η υποδομή και να πάψει η απομόνωση αυτών των απομονωμένων περιφερειών. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες αυτές. Θα δώσω τον λόγο στους συναδέλφους και θα παρακαλέσω πρώτα τον εισηγητή κύριο Βιδάλ Κουάδρας να λάβει τον λόγο. Αλλά προσοχή, μέχρι τις 4 πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση του θέματος, γιατί μετά έχουμε άλλα θέματα. Παρακαλώ όλοι λοιπόν συγκεντρώστε την προσοχή σας στα πλέον ουσιώδη για να προλάβουν όλοι να λάβουν τον λόγο. Ο κύριος Βιδάλ Κουάδρας. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Η μελέτη αυτή είναι χρήσιμο εργαλείο για να εξοικειωθεί κανείς με την παρούσα κατάσταση σε ό,τι αφορά τα δίκτυα διανομής ε, φυσικού αερίου και πετρελαιοειδών και πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι τα ισχυρά σημεία, τα ασθενή, προοπτικές για το μέλλον. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν ε, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τους συντάκτες της μελέτης και επιτρέπει σε κάποιον που δεν είναι εξοικειωμένος με το θέμα να πάρει γρήγορα μια γεύση, μια ε, ιδέα αρκετά πλήρη ε, του θέματος. Βέβαια, εμείς αυτή τη στιγμή μελετάμε ε, τον κανονισμό για την προμήθεια του φυσικού αερίου και της ασφάλειας μάλλον της προμήθειας και ε, όταν παραγγέλθηκε η μελέτη αυτή δεν είχαμε υπόψη μας τον κανονισμό αυτό και ε, κάποια ζητήματα όπως είναι το νήμιον 1 ή τα στρατηγικά αποθέματα, τα υπέρ και τα κατά δεν έχουν ληφθεί υπόψη ενδεχομένω όσο θα έπρεπε. Αν γινόταν τώρα η μελέτη θα ήταν πιο παρόντα, δεν θα υπήρχε αυτή η διαφορά φάσεως. Εν πάση περιπτώσει χρήσιμο είναι ως εργαλείο η μελέτη και ε, ευχαριστώ και συγχαίρω τους συντάκτες. Επιτρέψτε μου πρώτα να κάνω δύο ερωτήσεις. Μας είπαν αυτές τις μέρες, ακούμε, ότι οι υποδομές στο μεταφορό του φυσικού αερίου είναι ακριβά έργα και βαριά η επένδυση. Ε, μιλάμε εδώ για ε, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ μέχρι και δισεκατομμύρια. Αλλά όταν πρόκειται για τις στρατηγικές διασυνδέσεις και τη διεύρυνσή τους, για να υπάρχει και η δυνατότητα αντίστροφης ροής, δηλαδή να είναι διπλής κατεύθυνσης η ροή του αερίου, για να γίνουν αυτές οι βελτιώσεις, το κόστος είναι αρκετά περιορισμένο και βατό και προσιτό. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την αντίληψη που ακούγεται για να μπει η αντίστροφη ροή δηλαδή στους αγωγούς και στις στρατηγικές διασυνδέσεις είναι συγκρατημένο το κόστος και αν ναι, μπορείτε να μας δώσετε μια τάξη μεγέθους. Πόσο κοστίζει δηλαδή για να υπάρχει και αντίστροφη ροή στις ε, συνδέσεις που σήμερα δεν υπάρχει. Και η επόμενη ερώτηση αφορά τη διαχείριση της αγοράς. Πριν από 20 χρόνια το φυσικό αέριο ήταν στα χέρια μονοπωλίων, εθνικών. Με ένα και μόνο φορέα που είχε την αποκλειστικότητα, εισαγωγή, μεταφορά, διανομή, ε, αποθέματικα κτλ. Τώρα θεωρητικά έχει ανοίξει η αγορά, έχει απελευθερωθεί με κανόνες για την πρόσβαση ε, σε τρίτους. Έτσι λοιπόν ακούγονται διάφορες προτάσεις και κυκλοφορούν που λέγουν ότι ίσως να ήταν καλό να διαχειριζόμαστε με τρόπο ολοκληρωμένο ε, τη διαπραγμάτευσή μας και τη, τη συνδιαλλαγή μας με Κάποιου τρίτου εξωτερικούς προμηθευτές. Δηλαδή κάπου να συνεννοούμαστε. Και όταν αρχίζουμε τη διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές φυσικού αερίου, να μιλάμε όλοι με μία φωνή. Γιατί αυτό θα μας έδινε μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ. Σας ερωτώ ποια είναι η γνώμη σας για την πρόταση αυτή που ακούσαμε και πώς αξιολογείτε τη βιωσιμότητα και τη σκοπιμότητα μιας τέτοιας προσέγγισης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Καρβάιο. Thank um, Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτής της ε, έκθεσης. Εκτιμώ την εργασία σας, αλλά έχω μια ερώτηση που σχετίζεται με την παροχή στις απομακρυσμένες περιοχές. Εν συντομία, θίξατε το θέμα στην έκθεσή σας και πιστεύω ότι μια από τις λύσεις είναι οι αποθήκες LNG. Το θέμα είναι όμως ότι αυτό μπορεί να χρησιμεύσει σε περιοχές με ένα συγκεκριμένο όριο πληθυσμού. Έχετε σκεφτεί λύσεις, ε, για παράδειγμα, για τα νησιά με μικρότερους πληθυσμούς, όπως ε, ας πούμε, από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές, Αζόρες, Μαδέρα, λύσεις για νησιά με 350.000-150.000 κατοίκους. Έχετε ξεχτάσει τις πιθανές λύσεις για το υγροποιημένο φυσικό αέριο. μήπως είναι πιο εύκολο οι παράκτιες περιοχές της ε, Νορβηγίας να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα μικρότερα νησιά. Για την ώρα αυτές οι αποθήκες του υγροποιημένου φυσικού αερίου έχουν κατασκευαστεί για περιοχές με πληθυσμό πάνω των 500.000 ε, κατοίκων. Έχετε εξετάσει τις δυνατότητες για μικρότερους πληθυσμούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γιόρνταν Σίσελη. Eh, eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω κι εγώ μια ερώτηση για την υποδομή φυσικού αερίου. Μας είπατε ότι θα αυξηθεί η ζήτηση στο μέλλον. Επίσης και υπό το φως της κλιματικής αλλαγής. Μας δείξατε και ένα χάρτη όπου βλέπουμε διάφορα μελλοντικά έργα και σχέδια ανάπτυξης της υποδομής αγωγών φυσικού αερίου. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι να ακούσω την άποψή σας παρακαλώ για την επάρκεια αυτής της υποδομής. Δηλαδή θα μας φτάσει η μεγαλύτερη ζήτηση θα καλυφθεί από αυτά τα έργα ή θα χρειαστούν και νέα γιατί θέλει μεγαλύτερη ζήτηση. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να μάθω. Έχετε καθόλου στοιχεία για την αύξηση της ζήτησης φυσικού αερίου ανά κράτος μέλος. Και πώς συνδέεται αυτό με την υποδομή θέρμανσης και αν σκέφτεστε να δημιουργήσετε και νέα εργοστάσια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θεωρώ τη μελέτη αρκετά καλή αλλά θα ήθελα να θέσω μία πρώτη ερώτηση και γενική. Μας είπατε κύριε Πίτερσεν ότι τα μεγαλύτερα αποθέματα αερίου μέσα στο βελινεκές των αγωγών ή των υποπρόβλεψη αγωγών έχουν η Ρωσία, το Κατάρ, δεύτερο το Ιράν και μετά το Κατάρ. Αν δεν απατώμε, διεθνώς και έτσι είναι το ράνκιν των ε, προμηθευτών αερίου. Στη μελέτη όμως ε, δεν είδα να επικεντρώνεστε ούτε στη Ρωσία, ούτε στο Κατάρ, ούτε στο Ιράν ως μία πρόβλεψη. Όσον αφορά τη Ρωσία, ε, ήδη από ό,τι έχω καταλάβει με τον κύριο Πίμπαλξ και με την Επιτροπή και με στο Κοινοβούλιο, γιατί είμαι καινούργια βουλευτής, ε, υπάρχει πρόβλεψη η Ευρωπαϊκή η, Ένωση, η Κομισιόν να προχωρήσει σε μια εμπορική συμφωνία με τη Ρωσία, ε, η οποία θα είναι καθαρά εμπορική. Πουλάς, αγοράζω. Ε, και να αφήσουμε τα politics ε, ε, στην πάντα. Γι' αυτό λοιπόν θα περίμενα οι μελετητές να το είχαν κατά νου αυτό και να μας, κάπως να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την εμπορική μας σχέση με τη Ρωσία. Γιατί η Ρωσία είναι καθοριστική και ως προς το Ναμπούκο, δηλαδή το Ναμπούκο φαίνεται να μην είναι βιώσιμο. Από ό,τι ξέρω, γιατί δούλευα στην ενέργεια πριν από πολλά χρόνια, οι Αζέροι υπόσχονται σε όλους αέριο. Αέριο στο Ναμπούκο, αέριο στο South Stream κτλ. Αν δεν έχουμε διασφαλίσει τον προμηθευτή μας ότι μπορεί να μας διασφαλίσει 31 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου για τον Ναμπούκο ετησίως, δεν είναι βιώσιμος ο Ναμπούκο. Για να γίνει βιώσιμος ο Ναμπούκο θα πρέπει να μπουν ως μέτοχοι και οι Ρώσοι. Είναι μία σκέψη την οποία κάνω και γιατί, γιατί πέρυσι είχα δει τον εκπρόσωπο του State Department στα θέματα ενέργειας να λέει για τον Ναμπούκο ότι για να γίνει βιώσιμος κάπου πρέπει να έχουμε και τη Ρωσία. Η δεύτερη εναλλακτική που βγαίνει για τον Ναμπούκο είναι το Ιράν. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια πολιτική μάχη με το Ιράν στη Γενέβη. Από τη μία πλευρά βλέπουμε τα σάνξος να υπάρχουν, η Γερμανία και η Γαλλία πιέζουν. Από την άλλη πλευρά παρατηρούμε ότι η Αμερική τίνει και ένα χέρι έτσι κάπως συμφιλίωσης με το Ιράν. Δεν μπορούμε να αγνοούμε το Ιράν. Το Ιράν θα βοηθήσει πολύ, δεν ξέρω πώς θα πάει πολιτικά και τι θα γίνει, αλλά η μελέτη μπορεί να μας είχε δώσει κάποιο περίγραμμα τη σημασία του Ιράν και πώς μπορεί να βοηθήσει ε, <clears throat> το Ιράν ως προς την τροφοδοσία, ακόμα και τον Αμπούκο. Η χθεσινή συμφωνία Τουρκίας-Αρμενίας, μεταξύ πολλών άλλων, βλέπουμε εκεί και την Αρμενία ως χώρα διάλευσης από το Ιράκ και από το Ιράν. Ε, επικεντρώνομαι στο Νότο, γιατί η μελέτη ήταν πολύ καλή ως προς το Βορρά, αλλά βλέπω δυναμίες στο Νότο. Και πάμε ε, στην παράγραφο που έχετε για τη Μέση Ανατολή ε, και τον Αραβικό κόσμο. Ε, δεν συμφωνώ για την αναξιοπιστία που λέτε για τον Αραβικό κόσμο. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι των χωρών του Αραβικού κόσμου, το οποίο είναι πάρα πολύ αξιόπιστο στις ε, business που κάνουν και ιδιαίτερα οι χώρες του κόλπου. Εκεί ως προς το αέριο μας ενδιαφέρει το Κατάρ και το Μπαχρέιν πολύ αξιόπιστη συνεταίρη και θα έβλεπα πολύ καλύτερη την πρόβλεψη ενός αγωγού που θα μας προμήθευε αέριο από το Κατάρ και από τον Μπαχρέιν, εξαιρετικοί συνεργάτες σε όλα τους, από ό,τι σκέφτεστε από την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος δεν έχει αέριο τόσο πολύ όσο θα ε, ε μας ε, οδηγούσε σε μία τόσο μεγάλη επένδυση. Πέραν του γεγονότος, του γεγονότος ότι τα Εμμυράτα μπορούν και οι ίδιοι να επενδύσουν ως επενδυτές στον αγωγό. Μπορεί να μου πείτε οικονομικά πόσο βιώσιμο θα είναι, πόσο μακριά θα είναι. Αυτά είναι τεχνικές λεπτομέρειες. Αλλά όταν έχετε κυρίαρχες χώρες παροχής αερίου, τη Ρωσία, το Κατάρ και το Ιράν, δεν μπορεί να τις αγνοήσετε μέσα στη μελέτη σας. Έστω και αν φαίνονται εξωπραγματικές. Τα έχουμε δει ότι πολλά πράγματα γίνονται, παρότι μπορεί να μας φαίνονται ότι δεν γίνονται. Ε, και θα έλεγα ε, γενικά κύριε Πρόεδρε όσον αφορά το θέμα της ε, ενεργειακής ασφάλειας ότι διαπιστώνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο έχουν έτσι κάποια απόσταση από τον αραβικό κόσμο. Ε, απόσταση από τη Ρωσία που μας προμηθεύει θέλουμε να διαφοροποιηθούμε. Απόσταση από τον αραβικό κόσμο που έχουν ενέργεια. Ε, τότε πώς θα προχωρήσουμε προσπαθώ να καταλάβω. Ε, και θα έλεγα και κλείνοντας ότι πολλοί, πολλούς από τους αγωγούς που βλέπω στη μελέτη σας θα έπρεπε να σκεφτούμε σοβαρά να τους καταργήσουμε και να επικεντρωθούμε πώς θα συνδεθούμε με τις κυρίαρχες χώρες προμήθειας αερίου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριος Σέντσου. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την εισήγησή σας. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια και να υποβάλω μια ερώτηση για το σημείο 6-4 της παρουσίασής σας. Δηλαδή την διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου. Διότι είδα εδώ διάφορες πληροφορίες που οδηγούν στην ιδέα ότι δύο αγωγοί, το South Stream και ο Ναμπούκο, δεν μπορούν να τα κατασκευαστούν ταυτόχρονα γιατί θα είναι δύσκολο να βρεθούν ε, επενδυτές και για τους δύο αγωγούς ή αρκετό φυσικό αέριο για να τους προμηθεύει. Μπορεί να υπάρξουν κάποιες δυσκολίες όσον αφορά την ε, παροχή για ορισμένες χώρες μέλη για να να ολοκληρωθεί ο Ναμπούκο το 2015 ενώ το South Stream το 2013. Το συμπέρασμα δηλαδή είναι ότι θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε ένα μόνο ε, πρόγραμμα, δηλαδή το South Stream, διότι ε, εκεί υπάρχει και η χρηματοδότηση και η επαρκής προμήθεια σε φυσικό αέριο. Υπάρχει ένα φόρουμ για την ενέργεια στην Μαύρη Θάλασσα που έγινε στη Ρουμανία πριν δύο μέρες και ο πρόεδρος της εταιρείας ΕΝΗ ισχυρίστηκε ότι αυτά τα δύο προγράμματα δεν είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους αλλά παραπληρωματικά αλλά δέχτηκε πως η εκτιμόμενη χωρητικότητα του Ναμπούκο δεν αρκεί για να προμηθεύσει ολόκληρη την Ευρώπη με το φυσικό αέριο που χρειάζεται. Πρόσθεσε δε πως η ασφάλεια σε την ενέργεια παραμένει μεγάλο πρόβλημα, αλλά δεν είναι πλέον η πρώτη προτεραιότητα και ότι είναι απαραίτητο να διαφοροποιηθούν οι πηγές και να εφαρμοστούν και νέοι κανόνες. Αυτή είναι μια θέση την οποία εξέφρασαν και άλλοι αναλυτές και εμπειρογνώμονες στο τομέα. Όσον αφορά τον πολλαπλασιασμό των οδών μεταφοράς, των οδικών ε, Μάλλον, συγγνώμη, των, των τρόπων μεταφοράς, το South Stream μπορεί να είναι ε, μια εξασφάλιση. Εξαρτάται όμω, ποιε θα είναι οι βασικές πηγές προμήθειας φυσικού αερίου. Το βασικό πρόγραμμα τη Ένωση και κυρίω τη Κομισιόν και επίση πολύ σημαντικό για πολλά κράτη-μέλη είναι ο Ναμπούκο. Εν πάση περιπτώσει αυτό ίσχυε μέχρι τώρα. Και με βάση αυτό το ιστορικό, ποια είναι η άποψή σα σε σχέση με την επιλογή τη προτεραιότητα που θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με αυτά τα δύο προγράμματα. Ποιο από τα δύο προγράμματα θα πρέπει να θεωρηθεί προτεραιότητα εν ώψη της ανάγκης ε, διαφοροποίησης των πηγών φυσικού αερίου και της αύξησης της ασφάλειας σε ε, ανεφοδιασμό ενέργειας. Θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν οι μηχανισμοί ε, παρέμβασης εάν υπάρξει ενεργειακή κρίση και αν τα κράτη-μέλη αποφασίσουν να δώσουν προτεραιότητα στο πρόγραμμα South Stream. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. 10 Έχουμε ακόμη βέβαια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που επιθυμεί να σχολιάσει, αλλά και ο ίδιος ο κύριος Πέτερσεν της θα ήθελε να απαντήσει. Ο κύριος Βάγνερ. Θα είμαι σύντομος κύριε Πρόεδρε και θα προσπαθήσω να τηρήσω κατά το δυνατόν τον χρόνο μου. Εμένα πολύ ενδιαφέρον μου φάνηκε ε, αυτό που είπε ο εισηγητής. Γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα από αγωγούς φυσικού αερίου και από ε, πέτρελαγωγούς. Έμαθα πάντως σήμερα, αλλά ξέρω πολλά για τα κράτη και για το πώς λειτουργούν τα κράτη. Και τρομάζω λίγο όταν βλέπω πώς ε, όλα αυτά λειτουργούν στην Ευρώπη. Γιατί διαπιστώνω ότι υπάρχουν κράτη και κράτη πολύ όρημα παραλύουν όταν δεν έχουν φυσικό αέριο και υπάρχουν ιδιαίτερα βάρη και προβλήματα και για τις κοινωνίες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Από πλευράς θεωρίας ε, δημοσίων ε, εξουσιών και ε, διοικήσεων. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Και το πιο ενδιαφέρον από όλα όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη αυτό το διάστημα. Λοιπόν, τώρα έρχομαι στις ερωτήσεις μου σε ποιο βαθμό η σημερινή οικονομική κρίση και ε, η μείωση της ζήτησης σε ενέργεια που ε, συνεπάγεται, πώς αυτή μπορεί να επηρεάσει τα διάφορα έργα που γίνονται, ε, τις υποδομές. Γιατί στη χώρα μου υπάρχει μεγάλη διαμάχη στη δημόσια ζήτηση σχετικά με αυτό το θέμα. Γιατί έχει μειωθεί η ζήτηση και αυτό επηρεάζει έργα που τρέχουν και πολλές περιφέρειες της Ισπανίας. Επίσης θα ήθελα να τονίσω κάτι που είπε προηγουμένως ο συνάδελφός μου ο κύριος Βιντάλ άδρας για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα θέματα. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό το στοιχείο. Θα πρέπει να δώσουμε μια απάντηση. Ο Βιντάλ Άδρας μίλησε για κάποιο όμιλο αλλά θα μπορούσαμε να δούμε πρόσωπα δημοσίου δικαίου ε, και ιδιωτικού δικαίου, εμπορικές επιχειρήσεις ή κάτι αντίστοιχο για να ε, δώσουμε μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Ελπίζω να είμαι σύντομος όπως μα ζητάει πάντα ο πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Thank you so much. Mr. Correra de Campos. Thank you, Mr. Chairman. Obrigado, Sr. Presidente. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Correra de Κάμπος. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτήν την εισήγηση, αλλά να σας πω πως ε, επίσης, όπως και κάποιοι άλλοι από τους συναδέλφους, πως υπάρχει μια άλλη όψη της πραγματικότητας που δεν ε, μας την παρουσιάσατε. Και η άλλη όψη είναι ότι κοιτάμε μέσα στην Ευρώπη, αλλά δεν εξετάζουμε τις στρατηγικές εκείνων που είναι οι προμηθευτές μας. Τελευταίο παράδειγμα, η σημαντική συμφωνία Ρωσίας-Κίνας για παροχή ενέργειας για 20 χρόνια. Ποια είναι η σημασία αυτής της συμφωνίας ε, για τον δικό μας βασικό προμηθευτή, τη Ρωσία δηλαδή, που μας παρέχει το 30%. Ποια είναι η σημασία αυτής της συμφωνίας ε, στην συλλογική της παραγωγή και ποια είναι η δική μας ε, ε, διαπραγματευτική δύναμη. Τι αντιπροσωπεύει για μας αυτή η δυνατότητα αγοράς που έχουμε, η αγοραστική μας δύναμη. Θεωρώ πως η ερώτησή μου είναι γενικού ενδιαφέροντος, συγγνώμη που μακρηγόρησα, αλλά πιστεύω πως θα ωφελήσει όλους τους συναδέλφους. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέει ο Σας ευχαριστώ και εγώ για αυτή την πολύ λεπτομερή παρουσίαση. Και εφόσον δεν έχουμε τόσο χρόνο στη διάθεσή μα, θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή σε δύο ερωτήσει. Μιλήσαμε για την χρήση του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Αλλά δεν είδα καμιά σχέση με το CNG, δηλαδή το αέριο που είναι τεχνολογικά ως λιγότερο απαιτητικό και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε περιόδους κρίσης για μικρότερες περιοχές αλλά και επίσης για την αυτοκινητοβιομηχανία. Θα ήθελα να γνωρίζω λοιπόν αν το CNG θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά. Ενδιαφέρουσα τεχνολογία για μια τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή όπως η Ευρώπη. Και μια δεύτερη ερώτηση σε σχέση με αυτό που ήδη περάσαμε, δηλαδή την κρίση που είχαμε στις αρχές του χρόνου, όπου υπήρξε πρόβλημα με την ε, παροχή ε, τον Ιανουάριο μπορούμε να βρούμε μια κοινή λύση, μια κοινή διαδικασία για τη μετώπιση τέτοιων περιστάσεων στο μέλλον. Γιατί προφανώ είναι πολύ σημαντικό να δούμε, να έχουμε δηλαδή προγραμματισμένες λύσεις, προγραμματισμένη διανομή κτλ. Διαφοροποίηση. Ωστόσο θα πάρουν πολλά χρόνια. Θα περάσουν πολλά χρόνια μέχρι να υλοποιηθούν όλα αυτά. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε δυνητική κρίσιμη κατάσταση. Φυσικά δεν επιθυμώ καθόλου κάτι τέτοιο, το απεύχομαι, αλλά αν συμβεί κάτι παρόμοιο, τι θα κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε κάποιο διαπραγματευτικό πρόγραμμα, κάποια διαδικασία, είτε για να διαπραγματευτούμε τη Ρωσία, είτε με άλλους προμηθευτές. Ευχαριστώ. Ďakujem Σας ευχαριστώ. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν αναμένουμε να υπάρξουν προβλήματα στις προμήθειες αερίου για τα επόμενα χρόνια, τότε δεν θα αρκέσουν αυτά τα έργα διαφοροποίησης που προβλέπουμε. Συμφωνώ και με την κυρία Ζαβέλα, διότι για μας πολύ σημαντική θα αποδειχθεί η σχέση με την Ρωσία και βεβαίως οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Εξού και το ερώτημά μου προς εσάς. Είναι διατεθειμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει αποτελεσματικά σε μια προσπάθεια να απαλύνει και να διευκολύνει την ρύθμιση των σχέσεων των δύο αυτών χωρών και το ξεπέρασμα των διαφορών τους. Νομίζω ότι ορισμένε από τις ερωτήσεις θα τις απαντήσει καλύτερα η Κομισιόν, στην οποία θα δώσει ευθύ αμέσω το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και καλησπέρα σε όλους για αυτή την ενομερωτική έκθεση της COVID. Πιστεύω πως είναι μια πολύ καλή έκθεση που έρχεται μετά από την έκθεση τον Νοέμβριο του 2008 της ε, ανασκόπησης στρατηγικής για την ενέργεια καθώς και το πράσινο βιβλίο για τις ενεργειακές υποδομές. Όλα αυτά θα πρέπει να τα εξετάσουμε στο πλαίσιο ε, των μέσων για την μελλοντική ενεργειακή ασφάλεια που έχουν ήδη αναγγελθεί μέσω της ανασκόπησης της στρατηγικής για την ενέργεια. Ενεργειακή πολιτική θα είναι στο επίκεντρο της προσοχής των επόμενων χρόνων, όπως γνωρίζουμε όλοι, και έτσι αυτή η εργασία εντάσσεται πολύ καλά στις προπαρασκευαστικές μας ε, εργασίες. Υπάρχουν πολλά ζητήματα εδώ. Όπως γνωρίζουμε, όλες οι υποδομές αυτή τη στιγμή δεν αποτελούν ε, τμήμα των ε, διευρωπαϊκών δικτύων για την ενέργεια το πετρέλαιο μάλλον δεν αποτελεί τμήμα, ενώ το φυσικό αέριο είναι μέσα στα διευρωπαϊκά δίκτυα και ίσως είναι θέμα το οποίο θα πρέπει να το εντάξουμε στην ε, διευρωπαϊκή, στα διευρωπαϊκά δίκτυα για την ενέργεια. Ίσως λοιπόν αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε γιατί είναι ένα θέμα του να δούμε αν θα συνεχίσει να φτάνει το πετρέλαιο μέσω των αγωγών στην Ένωση ή μέσω των, ε, της ναυσιπλοείας, μέσω της Βαλτικής θάλασσας, του Εύξηνου Πόντου και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το θέμα του πετρελαίου. Είναι ανοιχτό το θέμα αυτό. Για το φυσικό αέριο τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Και η πολιτική που έχει ακολουθηθεί μέχρι στιγμής είναι ότι ευνοούμε όλες τις υποδομές που συγγενεύουν με τις υπάρχουσες διαδρομές και επιπλέον ε, αγωγούς που προμηθεύουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα και μέσα στο δίκτυο του 2006 για τις ενεργειακές κατευθυντήριες γραμμές που έχει οθετηθεί από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, έχουμε προγράμματα προτεραιότητας και προγράμματα κοινή ωφέλεια. Το Ναμπούκο είναι πρόγραμμα ευρωπαϊκού συμφέροντο, ενώ το South Stream, για παράδειγμα, τότε δεν ήταν μέσα στι κατευθυντήριε γραμμέ. Έχουμε λοιπόν ένα είδος ταξινόμησης αυτή τη στιγμή για τους αγωγούς φυσικού αερίου και φυσικά θα πρέπει όλα αυτά να τα αναθεωρήσουμε εν ώψη των νέων στοιχείων που προέκυψαν φέτος εν μέρη λόγω της ε, κρίσης ε, προμήθειας που είχαμε τον Ιανουάριο αλλά και λόγω των προσπαθειών που κάνουμε για να ενισχύσουμε την ασφάλεια ανεφοδιασμού όπως το σχέδιο προπολογισμού για την ασφάλεια προμήθειας ε, σε φυσικό αέριο που κατατέθηκε τον Ιούλιο. Σαφώς ε, η ασφάλεια σε ανεφοδιασμό εξαρτάται από την διαφοροποίηση των πηγών. Αυτό είναι σαφώς ο στόχος οποιασδήποτε πολιτικής, η διαφοροποίηση ε, διαδρομών και ε, προμηθευτών. Και γι' αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να καλύψουμε κάθε πιθανή πηγή φυσικού αερίου. Αναφέρθηκε το Ιράν, το Κατάρ, η Ρωσία. Βεβαίως και σήμερα παίρνουμε πάνω από το ίμιση των παγκοσμίων πόρων σε φυσικό αέριο και είναι σαφές ότι το να διευκολυνθεί η μεταφορά του φυσικού αερίου από όλες αυτές τις περιοχές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους στόχους μας. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τις δυνατότητες της Αφρικής ή της Νορβηγίας. Και φυσικά το υγροποιημένο φυσικό αέριο που διευκολύνει την μεταφορά φυσικού αερίου μέσω των πλοίων από ολόκληρο τον κόσμο. Το Μπάγκο, Αυστραλία, ε, που ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί πόροι, πολλές πηγές. Η ευρύτερη εικόνα λοιπόν είναι αυτή και οι αρχές είναι πολύ σημαντικές και επιπλέον φυσικά είναι πολύ σημαντικό να γίνεται ο κατάλληλος διάλογος ανάμεσα στην Ένωση που είναι ίσως πιθανότατα η καλύτερη αγορά στον κόσμο με 500 εκατομμύρια καταναλωτές που πληρώνουν πολύ καλές τιμές για την ενέργειά τους. Έχουμε δηλαδή ένα μέτρο ε, να αντισταθμίσουμε και να πετύχουμε τις καλύτερες συμφωνίες με τις χώρες προμηθευτές. Αλλά θα πρέπει να θυμίσουμε πως είναι οι εταιρείε που κάνουν τις συμφωνίες και αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε είναι να φτιάξουμε το σωστό ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε οι εταιρείε να μπορούν να προβαίνουν σε συμφωνίες που θα εξασφαλίζουν ασφάλεια και ε, ε, ασφάλεια νεφοδιασμού. Αυτό ε, είναι ο στόχος και το ερώτημα του κύριου Βιντάλκου, άντρα βεβαίω ήταν κέριο, ότι δηλαδή είναι πολύ σημαντικό για η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την ισχύ της ω εσωτερική αγορά 500 εκατομμυρίων καταναλωτών, ώστε να πετυχαίνει τις κατάλληλε συμφωνίες για τις εταιρείε τη, Όταν ε, έχει να συνομιλήσει με τη Ρωσία, το Κατάρ ή οποιοδήποτε πιθανό προμηθευτή. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναδώσω τώρα το λόγο στον κύριο Πέτερσεν για να απαντήσει. Σίγουρα δεν θα μπορέσετε να ανακαλύψετε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά μας πείτε για μερικά ζητήματα την άποψή σας. Έχετε το λόγο, κύριε Πέτερσεν. Ευχαριστώ. Σχετικά με την ερώτηση που έκανε πρώτος κύριος βουλευτή. έχει τα το δίκιο. Δεν είναι πολύ δαπανηρά τα συστήματα αντίστροφης ροής. Δεν είναι πάντα δυνατό να γίνει, αλλά κανονικά όταν υπάρχει αυτή η δυνατότητα δεν είναι πολύ ακριβή. Ε, σε ε, σχέση με τα θέματα αυτά των κρατικών μονοπωλίων, ε, είναι ένα ζήτημα που αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Uh, ε, το άλλο θέμα για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες και την ενδεχόμενη χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου ή συμπιεσμένου ενδεχομένως ε, μικρότερες ε, κοινότητες σε πιο αεροκατοικημένες περιοχές. Γνωρίζω ότι στην Ιαπωνία χρησιμοποιούν LNG και CNG για ανεφοδιασμό μικρών κοινοτήτων και απομακρυσμένων. Σίγουρα βεβαίως υπάρχει αυτή η δυνατότητα. ακριβή μεν η τεχνολογία, αλλά υπάρχει. Στη συνέχεια, νομίζω ήταν και άλλη ερώτηση. Σχετικά με τις προτεραιότητες του Ναμπούκο και του South Stream, ε, σας παραπέμπω και πάλι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι προτεραιότητα νομπούκο για τη διαφοροποίηση της ε, ε, γεωγραφικής κατανομής των προμηθευτών. Είναι πολύ ενδιαφέρον ο αγωγός Ναμπούκο. Και πώς επηρεάζει η ύφεση την ενεργειακή ζήτηση. Κανονικά θα περίμενε κανείς ότι με την ύφεση μειώνεται και η ζήτηση της ενέργειας. Τώρα, ανάλογα με τη διάρκεια της ύφεση ε, θα εξαρτηθεί ε, από αυτή η προσφορά και τα προβλήματα που έχουμε από την προσφορά. Oh, uh, Άλλη ερώτηση κατά πόσο αρκούν μακροπρόθεσμα οι παρούσες υποδομές για να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση της Ευρώπης σε φυσικό αέριο. Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς. Προσωπικά θα σας απαντούσα ότι τα έργα που είναι προγραμματισμένα μάλλον δεν θα φτάσουν, δεν θα είναι αρκετά. Εξαρτάται πώς θα αναπτυχθεί η αγορά του υγροποιημένου αερίου, κυρίως. Αλλά η σημερινή δομή των αγωγών φυσικού αερίου μακροπρόθεσμα δεν νομίζω να είναι αρκετή για τη ε, διανομή φυσικού αερίου σε όλη την Ευρώπη για να καλυφθεί η ζήτηση. Ε, Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές πηγές και τους προμηθευτές, απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και στην παρουσίασή μου και στο σημείωμα Δεν κάνουμε καμία αξιολόγηση για το κατά πόσο είναι σοβαροί όχι οι προμηθευτές αυτοί. Ε, όλοι είναι εμπορικοί εταίροι μας. Δεν υπήρχε ε, καμία αρνητική πρόθεση. Ε, αν κάτι τέτοιο φάνηκε δεν ήταν σκόπιμο πάνω στην παρουσίασή μας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χάνζεν και κύριε Πέτερσεν για την παρουσίαση της έκθεσής σας και της μελέτης και ε, την ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ και τους συναδέλφους για τις ερωτήσεις του. Και εδώ ολοκληρώνεται αυτό το σημείο της ημέρης της διάταξης και μπορούμε σε μισό λεπτό να ε, ανοίξουμε το επόμενο. Ευχαριστώ. It's very complicated, many questions. Terrible. Κυρίες και κύριοι, ας ε, προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε βέβαια ορισμένα τεχνικά προβλήματα, αλλά είναι μικρά και θα λυθούν γρήγορα. Η επιθυμία μας ήταν να ε, συζητήσουμε σήμερα τα της Ομάδας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών σε θέματα πυρηνικής ασφαλείας. Καλωσορίζω τον κύριο Στρέταρ. Καλώς ήρθατε. Τον Ιούλιο του 2009 υποβλήθηκε η πρώτη έκθεση, πρώτη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων σας και αυτήν θα μας παρουσιάσετε. Και έχουμε και τη δυνατότητα ευθύ αμέσω να μόλις δηλαδή περιοθεί η παρουσίαση να ε, συζητήσουμε μαζί σας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα αρχίσω μιλώντας σλοβενικά, έτσι θα αντιληφθείτε κι εσείς ότι είμαι σλοβένος, βεβαίως δεν ομιλώ εξ ονόματος της Σλοβενίας, είμαι επικεφαλής της ομάδας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών και αυτό θα ε, συνεχίζω στα αγγλικά. Ίσως με τον τρόπο αυτό να είναι και πιο εύκολη η συζήτηση ε, ε, μεταξύ μας. Η ENSREG που είναι και το ακρόνιμο της Ομάδας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών σε θέματα πυρηνικής ασφαλείας και κάπως τα, ε, βλέπω ότι οι διαφάνειές μου είναι λίγο πιο μικρές, ε, έχουν βγει λίγο πιο μικρές, αλλά τέλος πάντων από ό,τι ε, είχα προβλέψει στην αρχή. Πάντως Έχουμε στείλει, όπως ε, γνωρίζετε, την πρώτη μας ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά σε εσά και ε, θα μπορέσω να σας την εξηγήσω σήμερα. Θα καλύψω ε, ορισμένα θέματα. Θα αρχίσω με μια σύντομη παρουσίαση, διότι θεωρώ ότι οι πλοίονες εξημών δεν γνωρίζετε τόσο καλά τα θέματα ασφάλειας στην της πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη. Θα σας δείξω πρώτα τρεις διαφάνειες για να εξηγήσω ε, ποια ε, πράγματα αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε περίπου 150 εν λειτουργία πυρηνικούς αντιδραστήρες για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος σε 15 χώρες μέλη. Και παράγουν περίπου το 1 τρίτο όλου του ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι σημαντική ε, πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. Και βεβαίως πρέπει να πράξουμε πάνω το δυνατό ώστε η λειτουργία τους να είναι ασφαλής. Προσπάθησα εδώ να εξηγήσω ε, με ποιο τρόπο ε, εγγυόμεθα την ασφάλεια της πυρηνικής ενέργειας, όχι βέβαια μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παντού όπου χρησιμοποιείται τεχνικά θα ήταν εύκολο ή απλό να κατασκευάσει κανείς ένα πυρηνικό εργοστάσιο αν δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ασφάλεια. Επειδή όμως πρέπει, οφείλουμε να ε, τηρούμε τις ε, διατάξεις ασφαλείας, υπάρχουν πάρα πολλά συστήματα τα οποία προστατεύουν και ε, όλη την ασφάλεια του πυρηνικού εργοστασίου. Βάζουμε πρώτα ε, φορτώνουμε τη μεγαλύτερη ευθύνη σε αυτόν που χειρίζεται το εργοστάσιο. Πρωτίστως λοιπόν υπεύθυνο είναι αυτός. Σε κάθε λοιπόν τέτοιο εργοστάσιο έχουν πολλές, τέτοιο σταθμό έχουν πολλούς και περίπλοκους μηχανισμούς διασφάλισης ε, της ασφάλειας με ε, διάφορες διαδικασίες που προβλέπουν ακριβώς τι πρέπει να συμβεί για να είναι ε, για να υπάρχει ασφάλεια. Έχουμε και επάνω από αυτά τα εθνικά νομοθετικά και ρυθμιστικά συστήματα όπου ο νομοθέτης παρακολουθεί τι κάνει ο operator και αυτό βέβαια εξ ονόματος των, ιστόνομα μάλλον, του κυριαρχού λαού. Βέβαια αυτό ε, δεν αρκεί. Έχουμε και πίσω μας το κοινό, τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία παρακολουθούν με τεταμένη την προσοχή να δουν μήπως και κάτι δεν γίνεται σωστά ώστε να το καταστήσουν γνωστό και να το καταδικάσουν. Για να λειτουργήσουν σωστά οι εγκαταστάσεις μας πρέπει να τηρούμε αυστηρούς κανόνες. Πρώτα πρώτα ποια είναι τα φυσικά όρια. Ποιοι, πώς λειτουργεί η τεχνολογία, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από την χρήση της ποια είναι τα όρια εκείνα εντός των οποίων μπορεί να λειτουργήσει η εγκατάσταση. Το δείχνω γραφικά με αυτό το σχήμα, δηλαδή μπορεί, μπορούμε να κινούμεθα ανεξαρτήτως μέσα σε αυτό το πλαίσιο και να είμαστε πάντοτε ασφαλείς. Αλλά για να γίνουμε ακόμα ασφαλέστεροι βάζουμε και ε, νομικά πλαίσια. Το ευρωπαϊκό, μετά υφιστάμενο σε αυτό είναι το εθνικό, γιατί το ευρωπαϊκό δεν είναι πάρα πολύ ισχυρό. Έχουμε λοιπόν πολύ άκαμπτα εθνικά νομικά πλαίσια, τα οποία βασίζονται όλα σε διεθνείς προδιαγραφές και κυρίως της ε, ε Διεθνούς Αρχής Ατομικής Ασφαλείας, καθώς και άλλων διεθνών οργανισμών. Εκτός αυτού, κάθε νομοθέτης, κάθε ρυθμιστής δηλαδή, χορηγεί και την ε, έγκριση για τη λειτουργία, στενεύοντας ακόμη περισσότερο το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να κινείται η εγκατάσταση, ο σταθμός. Και εκτός αυτού, ο ίδιος ο operator θεσπίζει τις δικές του ακόμα πιο στενές διαδικασίες λειτουργίας. Άρα, εν τέλει, ο σταθμός πρέπει να είναι πάρα, πάρα πολύ προσεκτικός, ώστε να μην υπερβεί κάποια από τα πλαίσια αυτά και προκαλέσει κάποια κατάσταση ε, κινδύνου. Έρχομαι στην ιστορία της ΕΝΣΡΕΓ. Πρώτα, γνωρίζετε βέβαια ότι η πυρηνική ασφάλεια είναι καταρχήν εθνική ευθύνη, ότι κάθε χώρα η οποία διαθέτει πυρηνικούς σταθμούς έχει και έναν ε, πυρηνικό ρυθμιστή, ένα όργανο δηλαδή, το οποίο εντάσσεται στην δημόσια διοίκηση της εν λόγω χώρας και έχει ως ε, ρόλο να ρυθμίζει κανονιστικά τη λειτουργία των σταθμών αυτών. Οι εθνικές νομοθεσίες ακολουθούν τις ε, διεθνείς προδιαγραφές και είναι συνήθως αυστηρότερες. Είναι όμως σωστό επίσης ότι ποικίλουν από χώρα σε χώρα και κυρίως για λόγους ιστορικούς από το πώς εξελίχθηκε δηλαδή η πυρηνική ενέργεια σε διάφορες ε, χώρες. Υπάρχει και η συνθήκη Ευρατόμ που έχει η άνω των 50 ετών. Τότε βέβαια που ε, υπογράφτηκε η συνθήκη δεν θεωρούνταν τόσο σημαντικό το θέμα της πυρηνικής ασφάλειας και γι' αυτό έχει ε, αρκετά ευρύ χαρακτήρα η ε, συνθήκη εκείνη. Και από το καλοκαίρι που μας πέρασε έχουμε και νέο κανονισμό που είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για κάθε χώρα μέλος και απετέλεσε και το πρώτο βήμα προς ε, ένα, μια ευρωπαϊκή ρύθμιση. Τώρα, στο διεθνές σκηνικό. Κάθε χώρα που διαθέτει πυρηνική ενέργεια, ευρωπαϊκή δηλαδή, συμμετέχει και σε δύο σημαντικές συνθήκες. Η πρώτη είναι για την πυρηνική ασφάλεια και η δεύτερη είναι που είναι πολύ περιπλοκό το όνομά της δηλαδή και το βλέπετε από κάτω, είναι η ε, ε, συνθήκη για την ασφάλεια των ε, καταναλωμένων καυσίμων και την ασφάλεια των ραδιενεργών καταλήπων. Κάθε λοιπόν χώρα μέλος η οποία διαθέτει και όπου λειτουργούν στο εδαφός της πυρηνική σταθμή συμμετέχει και σε αυτές τις συνθήκες. Όπως είπα και προηγουμένως, η IAEA e διαθέτει προδιαγραφές, κώδικες και οδηγούς που επίση ακολουθούνται και υπό την αιγίδα του ΟΟΣΑ υπάρχει ενισχυμένη συνεργασία με έναν αριθμό επιτροπών οι οποίες ε, εγκύπτουν στα διάφορα θέματα σε διεθνές επίπεδο και έχουμε και την λεγόμενη ΟΕΝΡΑ που είναι ένα είδος λέσχης των ε, οργανισμών, των ρυθμιστικών οργανισμών. Λειτουργεί με τρόπο πολύ αποτελεσματικό. Με καλά αποτελέσματα. Έχουμε και τα λεγόμενα reference levels, επίπεδα αναφοράς, τα οποία είναι ένα είδος προδιαγραφών και τα οποία οφείλουν να σέβονται όλες οι χώρες. Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ιδέες για ένα κοινό πλαίσιο ασφάλειας έχουν ηλικία άνω των 10 ετών. Όμως το 2003 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει μια πρώτη προσπάθεια να εγκριθούν δύο οδηγίες, η μία για την ασφάλεια και η άλλη για ε, τα κατάλοιπα και δεν ήταν δυνατόν τότε βέβαια να εγκατέστη μάλλον δυνατόν να συμφωνήσουν όλες οι χώρες μέλη. Πέρασαν λοιπόν κάποια χρόνια με συζητήσεις και προδιετίας περίπου ιδρύθηκε η Επιτροπή για την ε, ε, ασφάλεια και την ασφάλεια των ε, ραδιενεργών καταλήπων και οι 27 χώρες μέλη έχουν διορίσει υψηλού επίπεδου ρυθμιστές που συμμετέχουν στην Εν Πρώτη φορά συνεδριάσαμε τον Οκτώβριο του 2007. Αρχικά κάναμε μια προσπάθεια να ξεκαθαρίσουμε ποιε είναι οι σχέσει μεταξύ χωρών μελών και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά αποφασίσαμε να λαμβάνουμε αποφάσει διασυνενέσεω. Καθορίσαμε του διαδικαστικού μα κανόνε, τον κανονισμό μα δηλαδή, και βάλαμε, καταστρώσαμε και τι προτεραιότητέ μα. Έχουμε, τα έχουμε βάλει όλα σε τρεις ε, ομάδες με τρεις βασικούς ε, τομείς. Πρώτα ε, τις ε, ρυθμίσεις για την ε, ασφάλεια, δεύτερον για τα καταναλωμένα καύσιμα και, το, τα ραδιενεργά κατάλοιπα και τρίτον ρυθμίσεις περί διαφάνειας που είπαμε από την αρχή ότι η διαφάνεια της εργασίας μας είναι ένα πρόβλημα. Ίσως καμιά φορά είμαστε αρκετά αδέξιοι σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το τι πράττουμε και αυτό πρέπει να βελτιωθεί. Έχουμε εργαστεί λοιπόν πάνω σε αυτούς τους στόχους ε, την τελευταία διετία και συνεχίζουμε. Τώρα, στην ομάδα εργασίας για την πυρηνική ασφάλεια που μιλήσαμε εκεί για πρώτη φορά για ένα ενδεχόμενο ευρωπαϊκό κανονισμό για τον τομέα της ε, πυρηνικής ασφάλειας, όπου υπήρχε από την αρχή μια διαφορά, μια διάσταση μεταξύ των χωρών της Ένωσης. χώρας χώρες ήταν υπέρ της οδηγίας, θεωρώντας ότι πρέπει να γίνει εναρμόνιση του τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είναι παράξενο που δεν υπάρχουν κοινοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τομέα αυτό, ότι Μπορεί έτσι να αποφευθεί κάποια επιδείνωση στον εθνικό τομέα, στους εθνικούς τομείς δηλαδή, και υπήρχαν και άλλοι, μεταξύ αυτών και εσεί, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή, που θα ήθελαν να γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχει και ένας μικρότερος αριθμός χωρών μελών που δεν επιθυμούν να υπάρξει τέτοια ρύθμιση. Με βασικό επιχείρημα ότι θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε η ευθύνη και την πυρηνική ασφάλεια να παραμείνει στο εθνικό επίπεδο και ότι θα ήθελαν να μπορούν να θεσπίζουν ακόμη αυστηρότερους κανόνες από αυτούς τους οποίους συμφωνούμε εδώ στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Εν τέλει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε σχέδιο νέας οδηγίας πριν από ένα χρόνο ακριβώς. Ακολούθησαν εντατικές συζητήσεις με ένα πρώτο, πάνω στο πρώτο σχέδιο δηλαδή και καταλήξαμε σε 10 βασικές αρχές οι οποίες θα πρέπει να περιληφθούν στην οδηγία. Θα σας τη διαβάσω σύντομα για να ε, προλάβουμε. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ε, βελτιώνουμε διαρκώς την πυρηνική ασφάλεια. Ποτέ δηλαδή δεν μπορούμε να αρκεστούμε σε κάτι που έχουμε επιτύχει. Πάντα πρέπει να προσπαθούμε περισσότερο. Δεύτερο, το δικαίωμα να επιβάλλονται αυστηρότερες ακόμα, ε, αυστηρότερες ακόμα απαιτήσεις πυρηνικής ασφάλειας. Αυτό θα πρέπει να διατηρηθεί από τις χώρες μέλη δεν θα πρέπει να γίνονται θεμελιώδεις αλλαγές στην βασική αρχή. Δηλαδή θα πρέπει ο εθνικός μεθυμιστής να παραμείνει ο βασικά υπεύθυνο. Το ίδιο και το επόμενο. Ο ρόλος δηλαδή του National Regulator πρέπει να ενισχυθεί. Δεν θα πρέπει να επεκταθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θα πρέπει να γίνει κάποιο είδος υπερρυθμιστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά θα πρέπει να παραμείνει μια πλατφόρμα που να μπορεί να προβλέψει και κάποιες αλλαγές. Το επόμενο είναι ότι δεν θα πρέπει να ε, γίνει κατακαιρματισμός των πόρων που χρειάζονται. Επίσης θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα από την συνθήκη της πυρηνικής ασφάλειας. Η επόμενη αρχή αφιερώνεται στις χώρες εκείνες οι οποίες δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν πυρηνική ασφάλεια. Όποιος λοιπόν δεν επιθυμεί μπορεί ασφαλώς να παραμείνει εκτός. Το ένα το σημείο είναι η διαφάνεια και το δέκατο είναι η ξεκάθαροι ρόλοι και ευθύνες οποιονδήποτε εμπλεκόμενων οργανισμών. Αυτές λοιπόν είναι οι δέκα βασικές αρχές, οι οποίες όλες περιλαμβάνονται στη νέα οδηγία του Συμβουλίου. Το επόμενο θέμα που ε, απασχόλησε την ε, υποομάδα πυρηνικής ασφάλειας ήταν το θέμα του benchmarking, Είπαμε λοιπόν ότι κάθε χώρα που διαθέτει πυρηνική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμμετέχει στο λεγόμενο IRRS, το σύστημα δηλαδή benchmarking και εσωτερικών ελέγχων μεταξύ των χωρών μελών υπό την αιγίδα της Διεθνούς Αρχής Πυρηνικής Ενέργειας, ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται κάθε έκτο έτος και ότι θα πρέπει να γίνονται και αυτοαξιολογήσεις. Και ο τρίτος τομέας που απασχόλησε αυτή την υποομάδα είναι η χρήση της συνθήκης πυρηνικής ασφάλειας. Κάθε τρίτο έτος, ε, τρία χρόνια δηλαδή, θα πρέπει να γίνεται μια συνάντηση των ε, συμβαλωμένων μερών, όπου κάθε χώρα μέλος θα πρέπει να ε, παρουσιάζει την δική της περίπτωση και οι άλλες χώρες θα μπορούν να σχολιάζουν ποια πράγματα είναι καλά, ποια όχι και τι προτείνουν για να διορθωθούν. Μετά από αυτήν την συζήτηση θα πρέπει να συζητούμε, να δούμε ποια είναι τα κοινά θέματα και να προσπαθούμε να εφαρμόζουμε τα μαθήματα, τα διδάγματα δηλαδή, σε όλες τις χώρες μέλη. Και μετά έχουμε και την δεύτερη ομάδα, την διαχείριση δηλαδή των ραδιενεργών καταλήπων, που εργάζονται σε τρεις κατευθύνσεις. Πρώτα, ότι κάθε χώρα μέλος, ανεξαρτήτως του αν έχει πυρηνική ασφάλεια ή όχι, πυρηνική ενέργεια ή όχι, θα πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα διαχείρισης ραδιενεργών καταλήπων. Ώστε κάθε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει μια ξεκάθαρη, ένα, μια ξεκα, για την διαχείριση των ραδιενεργών καταλήπων. Το ίδιο εδώ benchmarking και peer review, δηλαδή η αξιολόγηση μεταξύ των εταίρων. Είναι και, αυτή, είναι και αυτά σημαντικά και μέσα στα πλαίσια του IRRS και το ίδιο, όπως και η συνθήκη της επενδυτικής ε, ασφάλειας, τα αποτελέσματα ή τα διδάγματα από την χρήση της Joint Convention θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για κοινή εφαρμογή. Στα διάρκεια αυτών των δύο ετών το Συμβούλιο δέχθηκε υποστήριξη από την ομάδα μας για το ε, ψήφισμα που εξέρωσε. Στον τομέα της διαφάνειας δίνουμε τώρα πια την τελική μορφή σε μια πολύ εκτεταμένη ιστοσελίδα που διαθέτουμε για να παρουσιάσουμε τα θέματα πυρηνικής ασφάλειας στο κοινό με τρόπο όχι προκατηλημένο. Θα αρχίσει η χρήση της από τα τέλη του έτους, αλλά ήδη από τα τέλη του μηνός Οκτωβρίου θα υπάρχει η πρώτη ε, εφαρμογή στο χώρο αυτού και ταυτόχρονα και ο οδηγός καλών πρακτικών. Για το μέλλον θα συνεχίσουμε την εφαρμογή του προγραμματός μας, θα προσαρμόσουμε το πρόγραμμά μας και ανάλογα με τις εξελίξεις θέλουμε να παίξουμε έναν ρόλο στην εφαρμογή της οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια. Είμαστε ε, σε θέση να συμβουλεύσουμε τα ευρωπαϊκά όργανα για οποιοδήποτε μελλοντικέ πρωτοβουλίες. Θέλουμε να προχωρήσουμε και μια ευρεία συνδιάσκεψη για θέματα ρυθμιστικών διατάξεων για τα πυρηνικά και βεβαίως να ανταποκριθούμε με εύκαμπτο τρόπο σε οποιαδήποτε σχετική πρωτοβουλία. Τώρα στο τέλος έχω κρατήσει ορισμένες προσωπικές μου απόψεις σχετικά με το έργο μας των δύο τελευταίων ετών όπως και σε κάθε τομέα έχουμε στις κοινωνίες μας έχουμε τα επίσημα ε, νομικά συστήματα τα οποία έχουν ως στόχο την διατήρηση της τάξης αλλά είμαστε όλοι καθημερινοί άνθρωποι που ε, κινούμαστε και συναισθηματικά και ζούμε στον καθημερινό πραγματικό κόσμο και έχουμε ανάγκη να κατανοήσουμε οι μεν τους δε για να μπορέσουμε να βελτιωθούμε. Πιστεύουμε λοιπόν μέσα στα πλαίσια αυτά ότι ένστριγγα αποτελεί μια καλή πλατφόρμα και μια θετική πρωτοβουλία που μας αναγκάζει εμάς τους ρυθμιστές ή ε, τους υπεύθυνους για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη να καθίσουμε, να συνεννοηθούμε, να συνομιλήσουμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, μπορώ να σας πω ότι οι συνεδριάσεις μας ήδη τώρα που έχουμε συνεργαστεί επί δύο έτη έχουν γίνει πολύ ευκολότερες από ό,τι ήταν τον πρώτο χρόνο. Μπορούμε να κατανοήσουμε πολύ καλύτερα τι θέλουμε να επιτύχουμε και καταλήγουμε στη συνένεση πολύ συντομότερα. Και για το μέλλον είναι σημαντικό να γνωριζόμαστε, να κατανοούμε ή μεν τους δε, να γνωρίζουμε ποιες λύσεις δίνονται στις διάφορες χώρες και ούτω καθεξής. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας γνωρίζει πια και μας κατανοεί. Όλοι μαθαίνουμε από τις εμπειρίες των άλλων θεωρώ ότι η ρέγγ θα πρέπει να παραμείνει όπως είναι, δηλαδή μια πολύτιμη πλατφόρμα, ε, μια ε, τράπεζα εγκεφάλων, αν μπορώ να το πω έτσι, που έχει κρίσιμο ρόλο να παίξει για την χορήγηση συμβουλών σε άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε κάπως πιο ελεύθεροι από ότι είναι άλλα ε, θεσμικά όργανα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε επίσης ότι οι ευθύνε για την πυρηνική ασφάλεια θα πρέπει να παραμείνουν στο εθνικό επίπεδο στα χέρια εκείνων οι οποίοι βρίσκονται και συμβιώνουν με τους πυρηνικούς σταθμούς. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι είναι μέσα στα πράγματα πρέπει να φέρουν και την πρώτη ευθύνη. Η ανταλλαγή ωστόσο πρακτικών και ιδεών για την συνεχή βελτίωση πρέπει να ενθαρρύνεται. Αυτά ήταν όσα ήθελα να σας πω και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για να σας απαντήσω σε όποιες ερωτήσεις έχετε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σίτα, για την εκτενέστατη ενημέρωση. Σας ευχαριστώ ε, που μας εξιστορίσατε λίγο και πώς ε, εξελίχθηκε ε, η εργασία σας, γιατί φαίνεται ότι είναι μια ολόκληρη διαδικασία προοδευτική που προωθείτε εσείς και οι συναδελφοί σας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουν ζητήσει ήδη πρώτοι συνάδελφοι τον λόγο. Η συνάδελφος Γιώργαν Σίσελη πρώτη. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω αγγλικά τώρα, γιατί η διερμηνία την προηγούμενη φορά που μίλησα δεν ήταν αρκετά σωστή και ακριβής. Ευχαριστώ τον δόκτωρο στητα για την παρουσίασή του. Και δεν σε ευχαριστώ μόνο επειδή είσαι Σλοβαίνος, αλλά επειδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε πάρα πολύ ε, την ίδρυση αυτής της ομάδας των ρυθμιστικών αρχών και έλαβε υπόψη όχι μόνο την ανταγωνιστική τιμή αλλά και τα ευεργετήματα από την πυρηνική ενέργεια γιατί δεν παράγονται αέρια του θερμοκηπίου. Ε, θα αυξηθεί λοιπόν η χρήση πυρηνικής ενέργειας στο μέλλον και τώρα είναι η σωστή χρονική στιγμή για να δούμε τι θα κάνουμε νομοθετικά για να επιληφθούμε και των θεμάτων της πυρηνικής ασφάλειας. Δόκτωρ Στρίταρ, διάβασα επίσης ε, και την έκθεσή σας και κατανοώ ότι ο ρόλος της ομάδας σας είναι, πώς να το πω, συμβουλευτικός. Είστε ένα σώμα συμβουλευτικό ε, για το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από την παρουσίασή σας λοιπόν, τι είδα είπατε ότι αντιλαμβάνεστε το μελλοντικό σας ρόλο ε, μόνο από την πλευρά της υλοποίησης και της εφαρμογής λιμένων αποφάσεων. Σας ερωτώ λοιπόν κάτι άλλο εγώ τώρα. Τα δικά μας καθήκοντα ποια είναι ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των νομοθετών. Πού πιστεύετε ότι πρέπει εμείς να επικεντρωθούμε και πού χρειάζεται νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδιαίτερα θα σας, να σας ρωτήσω τι ε, πιστεύετε για τη χρηματοδότηση του παροπλισμού πυρηνικών εργοστασίων και της ε, επεξεργασίας πυρηνικών αποβλήτων. Τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση. Θα πρέπει να είναι εξάρτητη βεβαίως, αλλά πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι δεν θα επηρεάζεται ε, η χρηματοδότηση αυτή από εθνικές πολιτικές ή ακόμα και από ε, σχέδιο ιδιωτικών εταιριών. Και ελπίζουμε και τα κονδύλια να είναι διαθέσιμα όταν θα τα χρειαζόμαστε. Επόμενη ερώτηση. Επανειλημμένα αναφέρατε και κάποιες διεθνείς ε, συμφωνίες, συνθήκες μάλλον ε, και συμβάσεις ε, υπό την αιγίδα της υπηρεσίας της Βιέννης. Αλλά όλα αυτά δεν λειτουργούν στην ουσία. Αν σκεφτείτε τι γίνεται όχι μόνο στην Ινδία αλλά και στο, Ιράν και ζητήματα διάδοσης πυρηνικού υλικού Παγκοσμίω λοιπόν, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει, λαμβάνοντα υπόψη ότι βλέπουμε αναγέννηση πυρηνική ενέργεια σε άλλα μέρη του κόσμου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έξι συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Υποθέτω ότι μπορεί να κλείσει ο κατάλογος εδώ και θα παρακαλούσα τους συναδέλφους να είναι σύντομη και κάνουν και ακριβείς ερωτήσεις για να ακούσουμε πολλούς. Η κυρία Τζαβέλα παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Dr. σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετική η παρουσίασή σας και εκτιμώ πολύ τις προσωπικές σας απόψεις. Παίζει μεγάλο ρόλο να έχουμε τις προσωπικές απόψεις ενός ανθρώπου που έχει δουλέψει χρόνια στο αντικείμενό του. Ιδιαίτερα το σημείο 2 ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Μετά το ατύχημα στο Τσερνομπίλ παρατηρείται ένα κλείσιμο των ε, σχολών πανεπιστημίων οι οποίες παρήγαγαν εξειδικευμένους μηχανικούς σε θέματα πυρηνικής ενέργειας. Δηλαδή, αν δείτε τα μεγάλα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, σχολές ε, που λειτουργούσαν ε, δεκαετίες πριν έχουν κλείσει. Η ερώτησή μου είναι, έχετε εξακριβώσει έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στα θέματα πυρηνικής ενέργειας, γιατί αυτό αφορά οπωσδήποτε την ασφάλεια της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας. Το δεύτερο, η δεύτερη ερώτησή μου είναι η εξής. Υπάρχει μόνο μία εταιρεία σε όλο τον κόσμο, η Ιαπωνική, η οποία φτιάχνει αντιδραστήρες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα κτλ. Πριν από δύο χρόνια υπήρχε waiting list για τους αντιδραστήρες αυτής της εταιρείας. Δεν ξέρω αν επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, να πω το όνομα της εταιρείας. Μια Ιαπωνική εταιρεία είναι, η Mitsubishi είναι. Υπήρχε waiting list 25 χρόνια ε, για έναν αντιδραστήρα. Ε, δεν ξέρω τώρα μπορεί να, έχει γίνει το waiting list 20 χρόνια. Ε, αυτό πώς αντιμετωπίζεται, γιατί υπάρχουν χώρες οι οποίες διατείνονται ότι προχωρούν σε μια πενταετία ε, σε χρήση πυρηνικής ενέργειας. Ε, το θέμα της έλλειψης εμπειρογνωμοσύνης από ε, πλευράς βιομηχανικής κατασκευής δεν σας φοβίζει. Ευχαριστώ πολύ. Herr Kollege Balschow. Ο συνάδελφος Ευχαριστώ πολύ, λέει κύριος Μπάλσου. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε. Βλέπουμε ότι γίνεται πάρα πολύ σοβαρή δουλειά εκεί, στην ΕΝΣΡΕΚ. Πώς γίνεται εκεί η λήψη των αποφάσεων, πώς λαμβάνουν οι αποφάσεις. Ε, είναι συνενετική και τα μικρά κράτη έχουν ε, ίδια βαρύτητα στην ψήφο του, ίδια στάθμιση με τα μεγάλα κράτη, όπω επίση και χώρε που δεν έχουν πυρηνικά συμμετέχουν εξίσου με εκείνε που έχουν πυρηνικά. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Θέλω να πω κάτι άλλο εγώ τώρα. Ε, είναι και ζήτημα ευθύνης και αρμοδιοτήτων. Υπάρχουν μερικές αρμοδιότητες που ακούμε ότι θα πρέπει να παραμένουν σε εθνικό επίπεδο. Όλα αυτά ακούγονται πολύ ωραία και συμπαθή, αλλά εδώ υπάρχει μια αντίρρηση. Τα θέματα ασφαλείας δεν αφορούν ε, ένα κράτος και μόνο κάθε φορά, αφορούν όλες τις χώρες. Δεν υπάρχει πουθενά καμία ανάγκη να θεσπιστούν κεντρικοί κανόνες πανευρωπαϊκοί για την ασφάλεια. Ή ένας ευρωπαϊκός κανονισμός, για παράδειγμα, δεν θα μπορούσε να ε, αποφασιστεί. Για να μην έχουμε συγκρούσεις μεταξύ διαφόρων κρατών που χρησιμοποιούν, ας πούμε, πυρηνική ενέργεια και κρατών που δεν έχουν καθόλου πυρηνική ενέργεια. και ως διεθνής οργανισμός, επαρκή οργανισμός της Βιέννη, η διεθνή Επιτροπή ατομική Ενέργειας για να επιβάλλει τους ίδιους κανόνες παντού, που να τηρούνται και όλες. Θέλω να κάνω και μια ερώτηση για την εξασφάλιση του εφοδιασμού σε ενέργεια. Ακούμε πολλές φορές τους αντιπάλους πυρηνικής ενέργειας να ισχυρίζονται ότι δεν έχουμε αρκετό ουράνιο ή δεν υπάρχουν ε, αρκετά αυτές ε, μονάδες καυσίμου. Εσείς το έχετε μελετήσει, το ξέρει η ΕΝΣΡΕΚ, αυτό το ζήτημα. Έχετε κάνει καμία πρόβλεψη για την ασφάλεια ανεφοδιασμού και εκεί. Έχουμε αρκετή πρώτη ύλη ε, για να είναι εξασφαλισμένη αυτή η πηγή ενέργειας ε, μακροπρόθεσμα. Η κυρία Χάρμς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στα αγγλικά η κυρία ε, Χάρμς. Έχω τρεις ερωτήσεις. Για το ανθρώπινο δυναμικό ε, και ε, γενικότερα την κουλτούρα της ασφάλειας θα πρέπει λέει να μελετηθεί περισσότερο. Δεν το κατάλαβα αυτό. Τι είναι η κουλτούρα ασφάλειας, safety culture. Αυτό είναι τα τεράστια προβλήματα, ας πούμε, ε, που ακούσαμε από την ελβετική κυβέρνηση για το εργοστάσιο του Βάτενφαλ που ενδιαφέρει και τη Γερμανία. Επίσης παρακολουθείτε το ζήτημα των εργαζομένων σε πυρηνικά εργοστάσια στη Γαλλία, γιατί πριν από λίγες εβδομάδες βγήκαν στον τύπο και διαμαρτύρηθηκαν σοβαρά ε, για τις συνθήκες εργασίας τις οποίες είναι αναγκασμένοι να ε, εργάζονται και είπαν ότι αυτό ε, είναι κίνδυνος και για το ίδιο το εργοστάσιο. Και επίσης, στην προηγούμενη θητεία, λίγο πριν λήξει, αποφασίσαμε μερικά ε, θέματα και συγκεκριμένα ένα κανονισμό για κοινέ προδιαγραφές για πυρηνικά εργοστάσια στην Ευρώπη. και ακούσαμε ότι αυτό δεν αντανακλά ε, τη σημερινή, το σημερινό επίπεδο τεχνολογίας και επιστήμης. Εσείς τι λέτε, κυρίως για τα εργοστάσια που είναι στο, σχέδιο του, στο στάδιο συγγνώμη, του σχεδιασμού. Και μια ερώτηση για τη Γερμανία. Έχουμε πολλά προβλήματα με την υπόγεια ε, αποθήκευση ε, πυρηνικών αποβλήτων. Το συζητά αυτό η στη Γερμανία. Έχουμε για ένα σχέδιο εκτάκτου ανάγκης όταν υπάρξει σοβαρό πρόβλημα. Στην κάτω Σαξονία υπάρχει ένα τέτοιο θέμα μια περιοχή όπου θάβονται πυρηνικά απόβλητα και ενδεχομένω να μπορούσατε να το σκεφτείτε και πανευρωπαϊκά αυτό. Κύριος Οντή. Ε, Σα ευχαριστώ για την έκθεσή σα και για την παρουσίασή σα. Η πρώτη μου ερώτηση αφορά την ε, σύσταση τη δομή. σα. Αυτή τη στιγμή αποτελείται από του ε, διευθυντέ των ανεξάρτητων εθνικών αρχών και από εκπροσώπου τη Επιτροπή με παρατηρητέ την Ελβετία, την Ελβηγία, το Συμβούλιο και τη Γενική, την ε, Διεθνή Επιτροπή Ατομική Ενέργεια. Πιστεύετε ότι εδώ θα πρέπει να δημιουργηθεί κάποια κοινοβουλευτική δομή γιατί οι Ευρωπαίοι πολίτε ταυτόχρονα ανησυχούν για την πυρηνική ενέργεια αλλά ταυτόχρονα ε, κάποια κρατημέλη μπαίνουν στον πειρασμό. Κάποια κρατημέλη ε, άλλαξαν γνώμη εντωμεταξύ για αυτό το είδο την ενέργεια. Μήπως λοιπόν μια κοινοβουλευτική δομή σας φαίνεται ενδιαφέρουσα και επιταλέτε στη σελίδα 13 της εκθεσής σα ότι είστε ανεξάρτητοι. Αλλά Κατά την άποψή σας, ποια είναι η φύση και η σταθερότητα της ανεξαρτησίας σας, γιατί φαντάζομαι ότι ανήκετε στον δημόσιο τομέα της Σλοβενίας, ορίζεστε από την κυβέρνησή σας που έχει... Ε, δεν μπορεί να σας επηρεάσει, είστε πραγματικά ανεξάρτητος απέναντι στην κυβέρνησή σας και, και οι συνάδελφοί σας είναι ανεξάρτητοι, γιατί αυτό είναι αυτό που λέτε στην έκθεσή σας και όταν το διαβάζουμε και εμείς επιθυμούμε την ύπαρξη μιας ευρωπαϊκής αρχής που να είναι ανεξάρτητη. Και τελευταία ερώτηση. Ποιες κυρώσεις έχετε στη διάθεσή σας όταν υπάρχουν παρεκκλήσεις, όταν υπάρχει πούμε, ένα πρόβλημα ενός μεγάλου φορέα στην πυρηνική ενέργεια αυτή τη στιγμή που από ό,τι φαίνεται αποθηκεύει ε, απόβλητα, απόβλητα στο ύπεθρο στην Σιβηρία, τι ε, ενέργειες, τι ενέργειες προτίθεστε να προβείτε. Ο κύριος Μεστσάρος. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ τον κύριο Στρίταρ για αυτή την ε, πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, η παρουσίαση. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Στρίντερ πώς βλέπει την μελλοντική ανάπτυξη περαιτέρω εφαρμογής κανονισμών ασφάλειας στα πυρηνικά εργοστάσια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να υπάρχει μια αναλογία ανάμεσα στην ενέργεια που παράγεται και την περαιτέρω αύξηση του κόστους ασφάλειας και των άλλων του, υπόλοιπου κόστους. Ξέρω πως η ασφάλεια είναι το πιο σημαντικό, ωστόσο υπάρχει ένα ανώτατο όριο όταν είναι να, για, όπου μετά από εκεί δεν είναι πια, δεν αξίζει να παράγουμε τέτοιου είδους ενέργεια. Έχουν γίνει κάποιες τέτοιες μελέτες ή προγραμματίζονται τέτοιου είδους μελέτες για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Αναλογία δηλαδή κόστους ωφέλειας για την ασφάλεια. κυρία Ντατή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, η έκθεση που μας παρουσιάζεται σήμερα μας επιτρέπει να δούμε ποια είναι η κατάσταση προόδου όσον αφορά την εγγύηση μεγαλύτερης ασφάλειας της πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά, η παραγωγή της βερνικής ενέργειας δεν είναι πάντοτε συνενετική στην Ευρώπη. Βλέπουμε μάλιστα στη Γαλλία σε μια μεγάλη εφημερίδα εχθές μόλις ε, υπήρχε άρθρο για την διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων. Υπάρχουν διάφορες λοιπόν, διάφοροι προβληματισμοί, αλλά πιστεύω πως έχουμε κάθε την να κερδίσουμε από μια ασφαλή ε, και μετρημένη παραγωγή της ε, πυρηνικής ενέργειας. Στη Γαλλία ε, μας έχει βοηθήσει να έχουμε μεγάλη ανεξαρτησία σε ενέργεια, πράγμα το οποίο δεν είναι διόλο μελιτέο τη σήμερον ημέρα. Δεν είναι το μόνο πλεονέκτημα της πυρηνικής ενέργειας. Επιτρέπει, όπως είπε και ο πρώτος ε, συνάδελφος που παρενέβη, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Άρα λοιπόν ε, η πυρηνική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, πράγμα το οποίο έχουμε αποφασίσει μαζί στο πακέτο ενέργεια κλίμα το Δεκέμβριο του 2008 και επιπλέον επιτρέπει πολύ χαμηλότερες τιμές στην κατανάλωση. Η πυρηνική ενέργεια λοιπόν αξίζει τον κόπο να την ε, ε, εκμεταλλευτούμε. Ωστόσο, παρόλα αυτά τα πλονεκτήματα προκαλεί μεγάλες ανησυχίες σε θέματα ασφάλειας. Είναι κατανοητή αυτή η ανησυχία και γι' αυτό και διαρκώς επαγρυπνούμε. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ μεγάλες προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξάλλου απόδειξη όλων αυτών είναι η οδηγία για την ε, πυρηνική ασφάλεια που υιοθετήθηκε τον περασμένο Ιούνιο, που δείχνει την αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασφαλίσει την ολοένα και ασφαλέστερη ε, εκμετάλλευση της πυρηνικής ενέργειας. Η κατεργασία των ραδιενεργών αποβλήτων παραμένει θέμα. Η διαχείριση αυτών θα πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλιστεί. Θα ήθελα να χαιρετήσω την εργασία σας και να καλέσω σε τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν εθνικά προγράμματα για την ασφαλή διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων. Και πέρα από τα όσα ήδη αναφέρονται στην έκθεσή σας και τα όσα ακούσαμε απόψε, ε, θα ήταν δυνατόν να, κάνουμε μια κατα... να δούμε μια κατάσταση, μια, μια επισκόπηση της ε, κατάστασης στα διάφορα κράτη-μέλη. Όσον αφορά την μη τήρηση των κανόνων διαχείρισης των ε, ραδιενεργών αποβλήτων, ποιε είναι οι συστάσεις σας, τι θα πρέπει να γίνει ώστε τα κράτη-μέλη να φτάσουν στο βέλτιστο επίπεδο ασφάλειας. Υπάρχουν κάποιες νήξεις στην έκθεση, αλλά όχι λύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ο κύριος Ενά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας υποσχέθηκα να είμαι πολύ σύντομος και θα είμαι. Έχοντας ακούσει αυτά που μας είπατε μπορείτε να, να ισχυριστείτε ότι είναι αξιόπιστα τα πυρηνικά εργοστάσια στην Ευρώπη και αν ε, υπάρχουν διάφορα επίπεδα πώς κατατάσσονται και οι πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ε, θα πρέπει πανευρωπαϊκά να συγκεντρώσουμε τη γνώση μας ε, για την ασφάλεια, την πυρηνική, αλλά να μείνει στα χέρια της αγοράς. Μια σύντομη ερώτηση ο Παύλο Ρούμπιχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να πω ρητά ότι αυτά που έκαναν ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο κατόπιν παρενέσεως του ε, Κοινοβουλίου είναι υποδειγματικά. Και χαίρομαι που μπορούμε να κάνουμε και τέτοιες πρόοδους για αυτά τα θέματα τα πυρηνικά. Δεύτερον, γνωρίζουμε ότι η πυρηνική ασφάλεια είναι κάτι το οποίο θεωρούν απόλυτη προτεραιότητα και οι υπέρμαχοι και οι αντίπαλοι της πυρηνικής ενέργειας. Όλοι ε, είμαστε στην κατεύθυνση αυτή και ενδιαφερόμαστε να είναι στο επίκεντρο η ασφάλεια. Εγώ ε, θα ήθελα να μάθω ποια είναι τα βήματα που σχεδιάζετε αν βλέπετε ότι δεν τηρούνται ε, τα πρότυπα ασφαλείας. Η ΒΕΝΡΑ ή η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας τι κάνει ε, για να επιβληθούν αυτά τα πρότυπα. υπάρχουν κάποια εργαλεία επιβολής των μέτρων και τι σχεδιάζετε να κάνετε. Μάλιστα. Είχαμε κλείσει τον κατάλογο, αλλά πάρα πολύ σύντομα θέλει η κυρία Τσικάου να κάνει μια ερώτηση. Ελπίζω να συμφωνείτε. Υποθέτω ότι συμφωνείτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πολύ σύντομα να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Μιλάμε τώρα για αντιδραστήρες τετάρτης γενεάς. Με πολύ λιγότερα ε, απόβλητα. Ποιε είναι οι εξελίξει πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να μπορούμε στο μέλλον να μειώσουμε ακόμα περισσότερο ε, τα πυρηνικά απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγή αυτών των αντιδραστήρων. Ευχαριστώ. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λόγο τώρα έχει ο κύριος Φάρος. Σωστά το λέω. <clears throat> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μέλος της ομάδας NSREC και συνεπώς ε, φυσικά συμμερίζεται και τα όσα λέγει η έκθεση. Στην αλληλογραφία και με το Συμβούλιο και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο επίτροπός μου ε, διευκρίνησε ότι οι μελλοντικές εργασίες της ένστραξ στα πλαίσια της ασφάλειας είναι ευπρόσδεκτες, ιδιαίτερα μια εναρμονισμένη διαδικασία υποβολής εκθέσεων για να βελτιωθεί και η αξιολόγηση μεταξύ ίσων peer review και ο Επίτροπος μου τόνισε πόσο μεγάλη σημασία έχει για μας η διαφάνεια ε, αυτό ε, είναι ένα θέμα με το οποίο έχει ε, φορτιστεί η τρίτη ομάδα εργασίας στην ΕΣΡΕΚ και πολλά από τα θέματα που ανέφεραν οι βουλευτές έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι στο παρελθόν τα κανάλια, οι διάβλοι επικοινωνίες δεν ήταν όσο διαφανείς θα έπρεπε. Και τέλος θα να πω ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που η ΕΣΡΕΚ θα εξακολουθεί να εργάζεται και στο τομέα των αποβλήτων και με μεγάλη περιέργεια και ενδιαφέρον ε, περιμένουμε τις προτάσεις της ΕΣΡΕΚ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γνωρίζοντας ότι το Ευρωπαϊκό Πυρηνικό Φόρο που συνεδριάζει τη Βράγα και τη Βρατισλάβα συμμετέχει και εκείνο σε αυτή την προσπάθεια. Στα αγγλικά λέει κανείς είναι natural, με δύο λόγια δηλαδή υποστηρίζουμε την προσπάθεια αυτή. Κάνουμε και τη γραμματιακή υποστήριξη. Εμείς παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την υποστήριξη αυτή στην ΕΣΡΕΚ και θα προσπαθήσουμε να την ενθαρρύνουμε και να την εψυχώσουμε έτσι ώστε ε, να συνεχιστεί η καλή δουλειά και το η δεύτερη έκθεση είναι σαν την πρώτη. Ευχαριστώ κύριε Φάρος. Έχει ξανά το λόγο ο Δόκτωρ Στρίτερ. Πάρα πολλές ερωτήσεις. Well, ναι, όντω είναι πολλέ ερωτήσει. Ε, θα προσπαθήσω να απαντήσω στι περισσότερε. Θα ξεκινήσω από την αρχή. Ε, επιβλήθη μια ερώτηση σε σχέση με τα διενεργά κατάλοιπα και πώς αυτά μπορούμε να τα ε, διαχειριστούμε, αν μπορούμε να τα διαχειριστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αν υπάρχουν σχετικά κονδύλια. Πάντως σίγουρα ένα ταμείο διαχείρισης των διενεργών καταλήπων θα πρέπει να δημιουργηθεί έτσι ώστε τα παιδιά μας να μην χρειάζεται να χρησιμοποιούν τα δικά τους ταμεία για κάτι που χρησιμοποιούμε τώρα. Δηλαδή, θα ήταν ίσως σοφό λοιπόν κάτι τέτοιο να ε, ρυθμιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με την Σύμβαση για την Ασφάλεια της Πυρηνικής Ενέργειας και το θέμα της ε, χρησιμότητας ή της αποδοτικότητας, θα πρέπει να σας θυμίσω πως η Σύμβαση αυτή δεν σχετίζεται με τη μήνυ διάδοση των πυρηνικών όπλων και τα θέματα, το θέμα του Ιράν δεν έχει καμία σχέση. Ε, εμείς εδώ έχουμε να κάνουμε με κίνητρα δεν προβλέπονται κυρώσεις ε, για όσους ε, δεν πληρούν ε, τις συστάσεις, δεν τηρούν τις συστάσεις της σύμβασης, ωστόσο ε, ε, ε, αποτελούν μια πολύ μεγάλη επιρροή και δέχονται μεγάλες πιέσεις από τις άλλες χώρες όταν εξακριβωθεί πως κάτι δεν λειτουργεί σωστά σε κάθε χώρα. Και μπορώ να σας πω από την εμπειρία μου ότι είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να βελτιωθούμε. Όταν δηλαδή κανείς σε, σου λέει πως δεν το κάνει σωστά, τότε βελτιώνεσαι. τώρα, για το ειδικευμένο προσωπικό. Αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα, το γνωρίζουμε και προσπαθούμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, αναζητούμε λύσεις. Όταν λέω εμείς αναζητούμε, εννοούμε ολόκληρη το κλάδο της πυρηνικής ενέργειας, όχι βέβαια μόνο οι ρυθμιστές και οι επόπτες, αλλά πιστεύω πως αν καταφέρουμε να αλλάξουμε την γενική στάση απέναντι στην πυρηνική ενέργεια, ώστε να είναι πιο ρεαλιστικοί οι άνθρωποι απέναντι και όχι θετική. Είμαι πως και πάλι θα έρθει κόσμο σε, αυτήν, την, σε αυτόν τον κλάδο. Εδώ και δεκαετίες η πυρηνική ενέργεια έχει στιγματιστεί αρνητικά ε, στην ε, κοινωνία και δεν ελκύει τους νέους. Για μένα το βασικό που θα μπορούσε να αλλάξει την κατάσταση θα ήταν πραγματικά να αν αλλάξει η στάση απέναντι σε αυτόν τον κλάδο. Υπόθηκε πως οι ιαπωνικές ε, πυρηνικές κατάστασεις είναι καλύτερες. Εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ κάτι τέτοιο. Υπάρχουν πολύ λίγοι προμηθευτές ε, πυρηνικής ενέργειας σήμερα στην αγορά, 4-5. Ένας εξ αυτών είναι ευρωπαϊκός, ένας άλλος ε, αμερικάνικος και ο τρίτος ιαπωνικός και μετά έχουμε τη Ρωσία και την Κίνα που φτιάχνουν τα δικά τους ε, πυρηνικά εργοστάσια. Το πρόβλημα είναι η κατασκευή των ε, αντιδραστήρων και των ε, των αντιδραστήρων η Ιαπωνία μόνο είναι σε θέση τώρα να το κατασκευάσει, ε, γιατί όλες οι άλλες χώρες είχαν σταματήσει να κατασκευάζουν ε, εδώ και 20 χρόνια. Το Ιαπωνικό, ε, ο Ιάπωνας κατασκευαστής ήδη έχει κλείσει για τα επόμενα 15-20 χρόνια δουλειά. 25 χρόνια για την κατασκευή ενός αντιδραστήρα. Δεν είναι πολύ μακριά να σκεφτούμε την εισαγωγή μιας νέας εγκατάστασης. Οι διαδικασίες μας ε, για την έγκριση από περιβαλλοντική άποψη να πάρουμε όλες τις εγκρίσεις, λειτουργίες ε, σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο, είναι τόσο χρονοβόρος που όντω μπορεί να πάρει 25 χρόνια η ολοκλήρωση της κατασκευής και η έναρξη εφαρμογή του. Πράγμα το οποίο καθιστά αυτήν την πηγή ενέργειας πολύ υποδέστερη από άποψη ανταγωνισμού σε σχέση με τις άλλες. Το θέμα ενός κεντρικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό κάπως το έθεξα στην παρουσίασή μου και είπα πως δεν υπάρχει σαφή συνένεση για την ώρα. Υπάρχουν κάποιοι, και εγώ είμαι μεταξύ αυτών, που πιστεύουν ότι κάποιο είδος ε, ευρωπαϊκού κανονισμού, ένα κάποιο επίπεδο μάλλον κανονισμού θα ήταν υποφελές, ωστόσο υπάρχουν άλλοι που δεν θέλουν να υπάρχουν πολλά πολλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να έχουν τα χέρια τους ελεύθερα ώστε να κάνουν τους δικούς κανονισμούς σε εθνικό επίπεδο. Για την ασφάλεια σε προμήθεια δεν μπορώ να απαντήσω. Εμείς ασχολούμαστε μόνο με την ασφάλεια, όχι με την ε, εξασφάλιση ανεφοδιασμού. Και αυτό είναι θέμα άλλων και δεν μπορούμε να παρέμβουμε εκεί. Για... Τώρα, για τον ανθρώπινο παράγοντα και τα θέματα της ασφάλειας. Θα ήθελα να σας πω ότι ένας κακός οδηγός μπορεί να σκοτωθεί με το καλύτερο αυτοκίνητο, αν είναι αρκετά ανόητος ώστε να οδηγεί τρελά, ενώ ένας καλός ε, οδηγός μπορεί να οδηγήσει οποιοδήποτε αυτοκίνητο και να φτάσει ασφαλή στον, προορισμό του. Άρα λοιπόν ε, και ο ανθρώπινος παράγοντας και οι κανονισμοί ασφάλεια είναι εξαιρετικά σημαντικοί και πρέπει καθημερινά να τα αντιμετωπίζουμε ώστε να είμαστε ε, σε θέση να αναγνωρίσουμε όταν κάτι αναπτύσσεται προς την σωστή κατεύθυνση ή όχι. Γιατί όταν αναλύουμε κάποια καταστροφή, πάντοτε βλέπουμε ότι τελικά ήταν θέμα ανθρώπινου λάθους. Βασική πρόκληση λοιπόν για τον ρυθμιστή είναι να μπορεί να αναγνωρίσει αυτά τα πρώιμα στάδια επιδίνωσης. Γι' αυτό και θέλουμε να εξετάζουμε αυτά τα θέματα ακόμα πιο εις βάθος. Δύο ερωτήσεις ετέθησαν σε σχέση με κάτι που συνέβη στη Γαλλία πριν από λίγες εβδομάδες και το θέμα της ε, Γερμανίας, αλλά δεν νομίζω πως ε, δεν είναι το δικό μας ε, θέμα να μιλάμε για ειδικά προβλήματα οποιοδήποτε. Είμαστε περισσότερο σώμα συμβουλευτικό. Δεν ασχολούμαστε με, με μονομένες περιπτώσεις. Uh, should it be good to have somebody from Parliament in the in the answer? I don't know. Maybe it wouldn't be bad. Why not? Το αν θα ήταν καλό να έχουμε και κάποιον ε, από το κοινοβούλιο, στη... μάλλον να είχαμε ένα είδος κοινοβουλίου, γιατί όχι. Μαζί με, τη, με την Κομισιόν είμαστε 28, άμα είχαμε και κάποιον εκπρόσωπο του κοινοβουλίου, δεν ξέρω, δεν νομίζω να ήταν κακό, αλλά δεν ξέρω και αν θα ήταν και καλό. Σε σχέση με την ανεξαρτησία. Η ανεξαρτησία είναι κάτι που επαναλαμβάνεται διαρκώς. Αλλά η ουσία είναι ότι οι ρυθμιστές θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ανεξάρτητοι από τον κόσμο τον οποίον ελέγχουν. Αυτού δηλαδή που παράγουν την ενέργεια και την πουλάνε. Πρέπει να είμαστε ανεξάρτητοι, πρέπει να είμαστε στο ίδιο Υπουργείο, ούτε ε, ούτε στο ίδιο τμήμα, ούτε, εν πάση περιπτώσει, ό,τι αφορά την παραγωγή ηλεκτρισμού. Αλλά βέβαια είναι αδύνατο να πούμε ότι είμαστε απόλυτα ανεξάρτητοι από το καθένα. Είμαστε πάνω από την κοινωνία, είμαστε και εμεί τμήμα τη κοινωνία. Και οφείλουμε να ακολουθήσουμε τις κατευθύνσεις που δίνονται από την ίδια την κοινωνία. Πιθανές κυρώσεις τώρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα ως ένσρεκ. Το πολύ που μπορούμε να κάνουμε είναι πολύ χειρό ε, μήνυμα για κάποιες αντικανονικότητες που μπορεί να συμβούν, αλλά ελπίζω να μην χρειαστεί ποτέ να το κάνουμε. το θέμα του παζαρέματος, της, του, του, της ωφέλειας ανάμεσα στην παραγωγή και την ασφάλεια. Ποτέ δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι 100% ασφαλής. Γιατί την επο... μπορεί σε μια στιγμή να πέσει ένας μετεωρίτης πάνω στο κτίριο ή να πάνω σε ένα ε, πυρνικό αντιδραστήρα. Σε οποιοδήποτε είδος ανθρώπινης δραστηριότητας υπάρχει ένα επίπεδο εμπιστοσύνης ότι δηλαδή τα πράγματα θα λειτουργήσουν σωστά και ότι όντως τελικά αυτή η, η ζυγαριά γέρνει προς την θετική πλευρά. Τώρα, τι με ρωτήσατε, πώς μπορούμε να μειώσουμε το διοξίδιο του άνθρακα. Μα δεν είναι δική μας ευθύνη αυτό και δεν μπορώ να το απαντήσω. Και πάλι δεν μπορώ να κρίνω αν ένα πυρηνικό εργοστάσιο οποιοδήποτε είναι ασφαλέστερο ε, από κάποιο άλλο. Προσωπικά είμαι βέβαιος ότι ακόμα και το πιο άσχημα σχεδιασμένο πυρηνικό εργοστάσιο θα λειτουργεί σωστά αν είναι καλή η ομάδα ε, που το διαχειρίζεται. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες και μεταξύ αυτών ο ανθρώπινος παράγων είναι ο πιο σημαντικός. Το βασικότερο λοιπόν δεν είναι το πώς έχει σχεδιαστεί το εργοστάσιο, δεν είναι λόγος ανησυχίας. Πιο σημαντικό είναι να υπάρχει αυτή η κουλτούρα της ασφάλειας ε, στους εργαζομένους και στη συμπεριφορά τους. Και η επόμενη ερώτηση αντίστοιχη. τι θα γίνει αν δεν λαμβάνονται υπόψη διεθνεί προδιαγραφέ και πάλι. Εμεί δεν έχουμε, μάλλον να το πω αλλιώ ένδικα μέσα, δηλαδή έχουμε και δεν έχουμε. Η Βέρα έχει επίπεδα αναφορά και έχουμε δεσμευτεί όλοι ότι θα το μεταφέρουμε στην νομοθεσία μα. Μέχρι τέλη του έτου θα το κάνουμε στη Σλοβενία αυτό. Μέχρι τα τέλη του έτου τα επίπεδα αυτά αναφοράς θα είναι ε, υποχρεωτικά και θα επιβάλλονται δια νόμου στη Σλοβενία. Και είμαι βέβαιος ότι θα γίνει και στα υπόλοιπα μέλη τη μέρα αυτό αντιδραστήρε τέταρτης γενεάς και πώς προχωράει αυτό. Δεν είναι πάρα πολύ γρήγορη η πρόοδος, ε, το υπόσχονται μετά από 20 χρόνια κτλ. Δεν μπορούμε τώρα να βάλουμε ε, κανονιστικέ προδιαγραφές και απαιτήσει. Θα δούμε πώς θα αναπτυχθεί αυτή η τεχνολογία. Προς το παρόν τα πυρηνικά εργοστάσια που λειτουργούν σήμερα είναι με αντιδραστήρες ε, πίεσης ή ε, με βραστό νερό. Στη Σλοβενία έχουμε ένα εργοστάσιο που παράγει 40 κυβικά το χρόνο, που είναι το μέγεθος ενός γκαράζ, όχι περισσότερο. Αποβλήτων χαμηλής και μέσης ε, ενέργειας, ε, το, το καύσιμο είναι άλλη ιστορία. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χάρμς έχει ζητήσει πάλι τον λόγο. Μπορείτε να είστε σύντομοι. Για να αποφευθούν ενδεχόμενες παρανοήσεις, δεν είμαι βεβαίω ότι κατανόησα καλά προηγουμένως. Αν κατανόησα καλά, αυτό που είπατε ήταν ότι ο σχεδιασμός, το design ενός πυρηνικού αντιδραστήρως δεν είναι το κρίσιμο στοιχείο για την ασφάλειά του, αλλά το κρίσιμο για την ασφάλειά του είναι πώς γίνεται η διαχείριση του αντιδραστήρα. Αυτό με ενόχλησε κάπως, διότι και εδώ έχουμε συζητήσει και συζητούμε και εγκύπτουμε συχνά σε θέματα βελτίωσης της τεχνολογίας. Η τρίτη και τέταρτη γενεά των αντιδραστήρων έχει σημαντικά πλονεκτήματα. Παίζει ρόλο δηλαδή. Κατάλαβα καλά ή ο κ. Στρίταρ. Ε, βεβαίως δεν, πρόκειται, δεν θα έδινα εγώ ως ε, εθνικός ρυθμιστής έγκριση άδεια δηλαδή λειτουργία σε οποιοδήποτε αντιδραστήρα. Ασφαλώς το design παίζει σημαντικό ρόλο. Αλλά αυτό που είπα είναι ότι και πέραν του αρχικού design το σημαντικό στοιχείο είναι η ανθρώπινη διαχείριση, ο ανθρώπινος παράγοντας. Εσείς κατά πάσα πιθανότητα αναφέρεστε στους υφιστάμενους αντιδραστήρες στην Ευρώπη. Από όσα γνωρίζω όλοι η εν λειτουργία πυρηνική αντιδραστήρια στην Ευρώπη, από όποιον και αν έχουν χτιστεί στο παρελθόν, αναβαθμίζονται ώστε να φτάσουν στα επίπεδα που είναι αναγκαία σήμερα. Και επομένω από τη σημερινή σκοπιά μπορούμε να πούμε ότι είναι σχεδιασμένοι καλά. Βέβαια σήμερα δεν θα του σχεδιάζαμε έτσι. Είναι όμω σε αρκετά καλό επίπεδο σύμφωνα με τι γνώσει που έχουμε τώρα και εάν το συνδυάσουμε με το πώ λειτουργούν, πώ γίνεται η λειτουργία και η διαχείρισή του, μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Σας ευχαριστώ κύριε ε, Στρίταρ, δόκτωρ Στρίταρ, για τις πληροφορίες και για την σύντομη συζήτηση. Είμαι βέβαιος, άλλωστε το είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι θα μπορέσουμε να επανέλθουμε και θα σας παρακαλέσουμε ξανά να έρθετε εδώ να συζητήσετε μαζί μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Συνεχίζουμε αμέσως. Äh, Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, θα έρθω στο υπαριθμόν 5 θέμα, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Γεωσκόπησης. Η συγητής είναι ο κ. Γκράντε, ο οποίος δυστυχώ σήμερα κολλείεται. Αλλά βεβαίως ε, έχει στείλει εκπρόσωπό του την κυρία Γιούντιτ Μέρκες, που θα τον αντικαταστήσει, θαυμάσια, θα μας πει με λίγα λόγια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 Uh, uh, um, ε, μάλιστα. Ε, εκπροσωπώ εδώ, ε, αντικαθιστώ μάλλον τον Νόμπερτ Κλάντε που δυστυχώς κολλείται και μου ζήτησε να πω δύο λόγια για τις ερωτήσεις και τις εξελίξεις σχετικά με το πρόγραμμα τηλεπισκόπησης GMES. Uh, Μέχρι τώρα είναι ένα από τα πολύ ε, επιτυχημένα σχέδια. Βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια, είναι καθοδόν. Υπάρχουν μερικά προβλήματα προς επίλυση, διότι το GMS είναι πραγματικά καθοδόν, αλλά είναι ένα σχέδιο ερευνητικό που βαίνει προς το τέλος του. Έτσι λοιπόν ε, στο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα δεν υπάρχει δυνατότητα να έχουμε ε, λειτουργία. Δηλαδή το λειτουργικό ε, σκέλος δεν εντάσσεται σε αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα. Και τι γίνεται όταν τελειώνει μια έρευνα και σου χρειάζεται ένας δορυφόρο στο διάστημα για να τεθεί σε ισχύ αυτό. Χρειάζεται να υπάρχει ένας προϋπολογισμός για το λειτουργικό κόστος το οποίο αυτή τη στιγμή δεν καλύπτεται. Και θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξουν κονδύλια από το ερευνητικό πρόγραμμα. Είναι κονδύλια που ε, αφιερώνονται στην έρευνα αποκλειστικά και θα θέλαμε αυτά να μεταφερθούν και να καλύψουν ε, το λειτουργικό κόστος. Ένα τμήμα αυτών δηλαδή. Ένα τμήμα του προγράμματος και αυτό να χρησιμοποιηθεί και ως προηγούμενο, να αποτελέσει προηγούμενο για να αντληθούν τα κονδύλια για το πρόγραμμα GMS. E Στη συνέχεια υπάρχει και ένα ζήτημα, μια ερώτηση για τη χρηματοδότηση των δορυφόρων των ίδιων. Ήδη υπάρχουν ε, μερικοί δορυφόροι σε τροχιά, αλλά χρειαζόμαστε ε, χρηματοδότηση για να ολοκληρωθεί αυτό το πρόγραμμα και να είναι ε, έτοιμοι προς εκτόξευση οι δορυφόροι. Λοιπόν, πού θα βρεθούν τα κονδύλια για από εκεί, γιατί και αυτό δεν υπάγεται στο ε, ευρυντικό πρόγραμμα και κάπου πρέπει να βρούμε τα χρήματα αυτά. Μετά, και άλλη ερώτηση. Έχω τρεις βασικές ανησυχίες δηλαδή. πέρα από το γεγονός ότι πηγαίνει καλά αυτή η προσπάθεια, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, είναι σε τροχιά και γυρίζει ο δορυφόρος και λειτουργεί. Συλλέγει κάποια στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία θα παρέχονται δωρεάν. Δηλαδή, ένας οργανισμός που θέλει να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να πληρώνει ή θα έχει ελεύθερη πρόσβαση, δωρεάν πρόσβαση. Διότι εμείς θέλουμε να πετύχει αυτό το πρόγραμμα ε, GMES και για να τονωθεί και προωθηθεί η καινοτομία ε, υπάρχει αυτή η ιδέα να είναι δωρεάν η παροχή και να έχουν κοινή πρόσβαση και όλες οι εταιρείες και οι νέες και οι καινοτόμες. Και μια τελευταία ανησυχία αφορά το συντονισμό του προγράμματος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τεθεί σε λειτουργία το πρόγραμμα GMS. Ποιος θα το λειτουργεί, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Αυτή το κατασκευάζει. Ο συντονιστής ποιος θα είναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ποιος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων, άλλη Γενική Διεύθυνση. Αυτό το σημείο ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί. Και αν είναι όντως ο συντονιστής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε είναι κάλλιστα σε θέση να κάνει προγράμματα, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι ε, ένα θεσμικό όργανο που να έχει ως βασική αρμοδιότητα τη διαχείριση των προγραμμάτων. Και επειδή προέρχομαι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ ικανή Επιτροπή για άλλα θέματα, αλλά όχι για να διαχειρίζετε τέτοιου είδους προγράμματα. Λοιπόν, ποιος έχει το συντονισμό. Αυτά, βασικά. Είχε να πει ο συνάδελφος Νόμπερτ Γκλάντε και εγώ για να σχολιάσουμε το πρόγραμμα GMES. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Ντατή. Euh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν με το ναι του Ιρλανδικού Δημοψηφίσματος για τη Λισαβόνα καθώς και με την επικύρωση της Πολωνίας η έναρξη ισχύω φαίνεται πια να κοντεύει. Δεν μπορούμε παρά να είμαστε ευχαριστημένοι γιατί ε, θα γίνει αυτό το διάστημα μια κοινή αρμοδιότητα και η Ευρώπη θα μπορέσει πλήρω να παίξει το ρόλο τη ω διεθνή δύναμη. Σε προηγούμενη συνεδρία είχα ρωτήσει τον κύριο Βέσεμπεργκ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη δημιουργία μια αρχιτεκτονική για μόνιμη διαχείριση του προγράμματο ε, GMS. Θέλω να επανέλθω από αυτό, διότι πριν είναι ένα σημαντικό στοιχείο του προγράμματο πρέπει να διευκρινιστεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια ανακοίνωση του 12 η Νοεμβρίου είχε θελήσει τη δημιουργία ενό Συμβουλίου Εταίρων και είχε προβλέψει εκεί ένα ρόλο παροχής βοήθειας για την εφαρμογή αυτού του προγράμματος που θα, θα αποτελείται και από εκπροσώπους των κρατών μελών ε, και εκπροσώπους του GMES μέσω υποδομών που θα μπορούσε να συνεργαστεί με την Κομισιόν σε στενή συνεργασία. Η Κομισιόν βεβαίω αναλάβει το συντονισμό, ε, φαίνεται αυτό φυσιολογικό, συλλογικό συντονισμό, αλλά δεν θα μπορούσε να μην κάνει διάλογο με τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, η ευρωπαϊκή διαστημικός οργανισμός, διαστημικός οργανισμός θα πρέπει να συνδεθεί με κάποιο τρόπο σε αυτό το Συμβούλιο. Η Κομισιόν το θυμίζει και ίδια στην στον ανακοινοθέντη ότι η καλή εφαρμογή του προγράμματος ε, απαιτεί συνεργασία μεταξύ πολλών φορέων και στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό μία δομή απλής διαχείρισης ε, ορατής και αποδοτικής για την σωστή αρχική εφαρμογή του προγράμματος. Θα ήθελα επίσης να σας υποβάλω ένα άλλο θέμα το οποίο δεν είναι γεγραμμένο στην πρόταση κανονισμού, αλλά που μπορεί να χρειάζεται να θυγεί, είναι η, η ε, πιστοποίηση των στοιχείων που δίνονται από τις υποδομές που θα πλαισιώνουν αυτό το πρόγραμμα. Θέλουμε στοιχεία τα οποία είναι πάντοτε πιο αποτελεσματικά, όπως το πρότεινε και η Γαλλική Προεδρία, να σκεφτούμε τον ορισμό ενός νομικού πλαισίου που θα επιτρέπει την πιστοποίηση των στοιχείων που προκύπτουν από το πρόγραμμα GMES. Μπορούμε να τους δώσουμε και νομική ισχύ για να μπορούμε να χρησιμοποιηθούν, ας πούμε, σε διευθέτηση διαφορών και επίσης να μπορέσει το πρόγραμμα αυτό να συμβάλλει στην, ε, στην ε, επίλυση διαφορών ε, στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, ας πούμε, για ρήψη ρήπων στη θάλασσα. Ε, θα πρέπει να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το πρόγραμμα για το καλό, το όφελος των συμπολιτών μας, αλλά και με διαφάνεια και άρα και αποδοτικότητα του προγράμματος GMES. E Ευχαριστώ πολύ για τη συμπλήρωση αυτή. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί άλλο συνάδελφο δεν θέλει. Πιέρι. Ο κύριο Σαπιέρη και ελπίζω να το πρόφερε σωστά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. <laughs> μου Ταριέ. Είμαι επικεφαλής του γραφείου GMS e και από ε, τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας ε, έχω αναλάβει την ευθύνη αυτού του προγράμματος εξ ονόμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να επανέλθω στα τρία θέματα που αρχικά μας τοποθετήσατε και θα επιμείνω λίγο στο τρίτο ε, για το Συμβούλιο των Εταίρων που μόλις τέθη. Να θυμίσω, όπως είπατε κι εσείς, για πρώτη φορά το πρόγραμμα αυτό τηλεπισκόπησης ε, της γης ε, μπαίνει σε ένα κανονισμό για να δούμε τι θα γίνει και πώς ε, εντάσσεται αυτό στο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα. Θα δούμε λοιπόν πώς πρέπει να διοργανώσουμε τη δουλειά μας, να οργανώσουμε τους εταίρους και πώς ε, θα χρηματοδοτήσουμε για να εδραιωθεί το σύστημα. Γιατί ρωτήσαμε πολύ τους χρήστες στην προετοιμασία του προγράμματος τα τελευταία χρόνια και τι μας λέγουν. Ότι αυτή είναι η πρώτη τους προτεραιότητα. Να είναι σίγουροι, να είναι βέβαιοι ότι θα εδραιωθεί αυτή η πληροφόρηση για να μπορούν να υποφελούνται. Ε, τη συλλογική προσπάθεια τη ασφάλεια και του περιβάλλοντο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα αυτό είναι και από τα βασικά σημεία που μας ε, ζητάει και η ε, ναυπηγική ε, βιομηχανία. Μας λένε ότι δεν μπορούμε μάλλον η βιομηχανία που παράγει τους δορυφόρους και η βιομηχανία ε, που έχει αυτή τη διαστημική τεχνολογία θέλει να έχει μια εξασφάλιση ότι θα υπάρχει ε, διάρκεια, ε, θα είναι βέβαια αυτή και η δράση μακροπρόθεσμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχει μια κοινοτική υπεραξία αποδεδειγμένη όμως με συνεχή παρακολούθηση και ε, αξιοποίηση και εκμετάλλευση των ε, δεδομένων για να είναι και χρηστικά αυτά από τις διάφορες κατηγορίες ε, χρηστών. Τώρα, για τη χρηματοδότηση βλέπετε νέα χρηματοδότηση με καλή κατανομή η παρατήρηση από το διάστημα, η παρατήρηση in situ, επιτόπου, όχι από το διάστημα, ανάπτυξη υπηρεσιών και user up που λέγεται αυτό στα αγγλικά, δηλαδή μια δράση, μια προετοιμασία όλων αυτών ε, των δεδομένων ε, εις όφελος ε, των χρηστών, γιατί πρόκειται για μια κοινοτική δημόσια επένδυση. Και θα πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση και έχει γίνει φυσικά η συζήτηση εδώ ε, μεταξύ των συνομοθετών και θα πρέπει να δούμε την ε, κατάλληλη ισορροπία και πώς θα κατανεμηθούν τα χρήματα αυτά στις διάφορες κατηγορίες και άξονες ε, του προγράμματος. Το δεύτερο, η πολιτική των δεδομένων, δηλαδή πώς θα παρέχονται αυτά τα δεδομένα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το συζήτησε αυτό το θέμα επανειλημμένος και συγκεκριμένα στα πλαίσια ε, του Συμβουλίου Υπουργών Αρμόδιων για το Διάστημα και πρότεινε κάτι άλλο που συνάδει πλήρως με αυτά που διεθνώς είχαμε ε, συμφωνήσει για την ε, ε, γεωσκόπηση, η πρόσβαση να είναι ως εξή. Την υποδομή αυτή θυμίζω ότι την έχουμε επομιστεί εμείς και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διασύματος. Οι άδειε λοιπόν για την πρόσβαση στα δεδομένα θα πρέπει να είναι δωρεάν, γιατί είναι δημόσια επένδυση. Έχουμε κάνει και μελέτες και αν θέλουμε να ε, αναπτυχθεί αυτός ο κλάδος και να είναι χρήσιμο και καινοτόμο αυτό το πρόγραμμα υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι δωρεάν γιατί πάρα πολλέ μικρομεσαίες επιχείρησεις ενδιαφέρονται να βρουν κάποια είσοδο σε αυτή την αγορά. Το τρίτο που αναφέρεται για την οργάνωση των εταίρων, μιλήσατε για το συντονισμό του προγράμματος. και το Συμβούλιο των Εταίρων, θέλω να θυμίσω την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2008 που προσπάθησε να παρουσιάσει τις μεγάλες κατευθυντήριες γραμμές της διαχείρισης του προγράμματος ΖΕΜΕΣ. Από την πείρα μας γνωρίζουμε, έχουμε διδαχθεί και προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι γενικό συντονιστής για το πώς θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα και σε ό,τι αφορά τα τεχνικά θέματα της εφαρμογής και διαχείρισης να βασιστούμε σε δομές που ήδη υπάρχουν στην Ευρώπη. Από την αρχή το Συμβούλιο μας έβαλε δύο προσανατολισμούς. Πρώτον, να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες των χρηστών και το δεύτερο να αξιοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα τις υπάρχουσες σήμερα δυνατότητες στην Ευρώπη δεν μας ενδιαφέρει εμά να έχουμε επικαλύψεις ό,τι υπάρχει να μεταφερθεί και σε κοινοτικό επίπεδο. Γι' αυτό το δεύτερο λοιπόν προτείνουμε να βασιστούμε σε υπάρχοντες οργανισμούς που ασχολούνται με αυτά τα θέματα τηλεπισκόπησης, γεωεπισκόπησης ε, και είναι η UMETSAT που είναι η μετρολογική δορυφόροι και λειτουργούν ήδη σε ό,τι αφορά τη συστηματική ε, παρακολούθηση και ε, στο μεταξύ ενδιάμεσα για άλλου είδους ε, παρατήρηση η ΕΣΑ, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, αναμένοντας ένα νέο πλαίσιο για να εδρεωθεί μακροπρόθεσμα αυτή η υποδομή. Σε ό,τι αφορά τώρα το Συμβούλιο των Εταίρων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε ότι πέρα από την Ένωση και τη δική μας δραστηριότητα ε, θα άξιζαν και άλλες προσπάθειες να συντονιστούν. Προσπάθειες πάντα παρατήρησης της γης από το διάστημα. Θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει και αυτό ένας ανοιχτός συντονισμός με τα κράτη-μέλη και... Μας ενδιαφέρει πολύ η συζήτηση που γίνεται εδώ σε επίπεδο νομοθετών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε το εξή χρονοδιάγραμμα συμφωνήσει. Ανταλλαγή απόψεων στις 10 Νοεμβρίου, ενδεχομένω 2-3 Δεκεμβρίου συζήτηση, 10 Δεκεμβρίου προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 27-28 ε, συζήτηση και 4 Φεβρουαρίου στην Επιτροπή. Συμφωνείτε? Ωραία. Το επόμενο θέμα το έχουμε ξανασυζητήσει. Είναι δομέ διαχείριση για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορική ραδιοπλοήγηση. Ο κύριο Τωσενόφσκι είναι εισηγητή. Ε, θα μιλήσει πρώτα εκείνο και μετά κάποιοι άλλοι συνάδελφοι που θα ζητήσουν το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζω ότι έχουμε μια ελαφρά πίεση χρόνου και θα είμαι σύντομος, γιατί όντως το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό το θέμα, δεν είναι η πρώτη φορά που μας απασχολεί. Δομέ διαχείριση λέει για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης. Περί τίνος πρόκειται. Είναι τεχνική εναρμόνιση δύο προδιαγραφών. Είναι δύο οδηγίε. 1321 του 2004 και 638 του 2008. Χρειάζεται όμως αυτός ο συντονισμός, αυτή η τεχνική ρύθμιση, διότι έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές. Γνωρίζετε ότι και το ίδιο το πρόγραμμα Γαλιλαίος έχει ε, περάσει μεγάλες αλλαγές. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι η ασφάλεια του όλου συστήματος και είναι κρίσιμο και αποφασιστικό. Ενδεχομένω μπορεί να υπάρξουν και αλλαγέ του ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, του διαχειριστικού φορέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μεγάλη ευθύνη τώρα γιατί προετοιμάζει το όλο σύστημα και γι' αυτό το λόγο έχουν κατατεθεί και κάποιες τροπολογίες. θα πρέπει να ενισχυθεί η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Διοικητικό Συμβούλιο και από πλευράς ψήφων. Θα πρέπει να έχει το ίμιση των ψήφων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια αυτό ακόμα δεν έχει λήξει. Είναι ένα θέμα που είναι υποσυζήτηση. Ξέρω ότι τα θέματα αυτά είναι λεπτά. Η πρόταση επίσης ε, είναι ευαίσθητη. Θα μπορούσε να μας πει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θέση έχει. Εάν συμφωνεί με την άποψη αυτή ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στο Εποπτικό Συμβούλιο αυτού του οργανισμού θα πρέπει να κυριαρχεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη συνέχεια, διορίζει το Κοινοβούλιο στο όργανο αυτό και δικό του εκπρόσωπο, βέβαια με καθεστώς απλού παρατηρητή, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Και αυτό όμως είναι λίγο προβληματικό και περίπλοκο. Τι θα πει, ρόλος παρατηρητή. Δεν έχουμε καθόλου ενεργή συμμετοχή με αυτόν τον τρόπο ως κοινοβούλιο. Αλλά επειδή είναι τόσο σημαντικά τα θέματα αυτά, καλό είναι να συμμετέχει και το Κοινοβούλιο. Επίσης ζητούμε ανεξάρτητο οργανισμό πιστοποίησης, διαπίστευσης, ανεξάρτητο επαναλαμβάνω, γιατί τα θέματα ασφαλείας είναι πολύ σημαντικά για να εξασφαλίζει σε όλα τα κράτη-μέλη την ασφάλεια του συστήματος. Θα πρέπει λοιπόν να είναι πολύ υψηλού επιπέδου η ασφάλεια και να έχουν και διαπίστευση ασφαλείας ε, οι υπάλληλοι. Ξέρουμε ότι εδώ δημιουργούνται πολλά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ε, γι' αυτό χρειάζεται συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να ξεκαθαριστεί το θέμα της συμμετοχής της ε, στο υποπτικό Συμβούλιο και με τη στάθμιση και το θέμα της ασφαλείας είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα δύο για ένα σύστημα τόσο περίπλοκο. Θα σταματήσω εδώ γιατί την έχουμε ξανασυζητήσει, είπαμε αυτή την πρόταση. Θα ήθελα να ακούσω και τους συναδέλφους. Αλλά το θέμα αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ κρίσιμο και πάρα πολύ σημαντικό. Και τώρα που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 50% και πλέον είναι πολύ σημαντικό. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρούμπιχ πρώτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Εκπροσωπώ εδώ τη συνάδελφό μου την κυρία Νίμπλε, αξιότιμη συναδελφή του τελευταίου μήνες και χρόνια, εμείς οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ασχοληθήκαμε εντατικά με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Γαλιλαίο το Απρίλιο του 2008 μετά από πολλές αλλαγές και σκληρές διαπραγματεύσεις δόθηκε επιτέλους το πράσινο φως. Ωστόσο παραμένουν ανοιχτά ορισμένα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το μέλλον ε, του συστήματος ραδιοπλοήγησης με δορυφόρο. Μας χρειάζεται ο Γαλιλαίος ως ανεξάρτητο σύστημα ραδιοπλοήγησης, ευρωπαϊκό, και είμαι απαθήτατα πεπισμένη γι' αυτό, λέει η κυρία Νίβλερ, για ε, του κυρίου Ρίμπιχ. Αλλά όλα αυτά θα πρέπει να ε, έχουν ισχυρή βάση. Το θέμα δεν είναι να κάνουμε ένα σχεδιασμό μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το πρόγραμμα Γαλιλαίος. Από εκεί και πέρα τι γίνεται από το 2013 και μετά τι ως είναι. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες και οι ευθύνε θα πρέπει μακροπρόθεσμα να είναι ε, δεδομένες και γνωστές για να ε, μπορούν όλοι να κανονίσουν την πορεία τους. Επιπλέον θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό που ζητάει πάει για το Κοινοβούλιο, η διαφάνεια δηλαδή, να είναι δεδομένη και στο μέλλον. Και τελικά γιατί σε τελική ανάλυση το πρόγραμμα αυτό το χρηματοδοτούν οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι και δικαιούνται να γνωρίζουν τι γίνεται με τα χρήματά τους και να είναι χρηστή η διαχείριση. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει ε, να ενημερώνονται τακτικά για το πρόγραμμα, την πορεία του και τη χρησιμότητά του. Και μόνο έτσι μπορούν να ε, δικαιολογήσουν και το κόστο τους. Επιπλέον θα πρέπει να δούμε και ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Διοικητικό Συμβούλιο ε, της υπηρεσίας ε, GNSS. Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα αυτό που έχει σημασία είναι να τηρήσουμε το φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα και να μην επιτρέψουμε καμία ε, ολιγορία περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ρούμπιχ, στο παρόν δεν βλέπω κανέναν. Α, τον κύριο Ντί βλέπω. Πολύ σύντομα, ε, στη σελίδα 19, μια παρατήρηση λέει ότι το ελεκτικό συνέδριο εγκρίνει τους λογαριασμούς. Κοιτάξτε, βασικά τους ελέγχει το ελεκτικό συνέδριο, δεν τους εγκρίνει τους λογαριασμούς. Θα κάνω τροπολογία προς την κατέση αυτή. Ευχαριστώ για την υπόδειξη. Äh, Κύριος Καραμίτσος έχει το λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Yes, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για την υποστήριξή του προς την πρόταση, πώς θα προχωρήσουμε. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα που τα έχουμε συζητήσει την περασμένη φορά. Επιτρέψτε μου να επαναλάβω μερικά για να διευκολύνει αυτό τη σκέψη σας για τα επόμενα στάδια. Ποια είναι η βάση της πρότασής μας. Αυτή η βάση ήταν ο κανονισμός του 2007, ο 683, που πραγματικά δημιουργεί, μάλλον ορίζει το ρόλο της Κομισιόν, το ρόλο του GSA, γιατί Επίτα προχωρά για το πώς θα πρέπει να γίνονται οι προμήθειες και όλες οι διαδικασίες. Εμείς ε, ζητήσαμε την ενίσχυση του ρόλου της Κομισιόν στο Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο του GC, γιατί από τη στιγμή που αποφασίστηκε πως η Κομισιόν είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του προγράμματος, θα έπρεπε να έχουμε και τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση και δεν μπορούμε να είμαστε σε μια κατάσταση όπου στο Συμβούλιο ας πούμε, θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του συστήματος ασφαλείας να μην λαμβάνεται υπόψη η Κομισιόν, γιατί είναι υπεύθυνη. Υπεύθυνη για τις ευθύνες. για τη συνολική ασφάλεια και μετά δεν μπορεί να είναι δηλαδή εκείνη υπεύθυνη για την ασφάλεια και μετά να λαμβάνονται οι αποφάσεις από κάποιο άλλο όργανο στο οποίο δεν συμμετέχει καν. Γι' αυτό και θέλαμε η Κομισιόν να συμμεριστεί αυτή την ευθύνη. Αν θέλει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να είναι υπεύθυνοι για κάτι, θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι ε, εφόλες της ύλης. Επίσης πιστεύουμε ότι είναι εξίσου σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει κάποιο ρόλο, ακόμα και αν είναι ένα μικρό ρόλο, να είναι να συμμετέχει στο Συνδικητικό Συμβούλιο. Διότι και πάλι ο κανονισμό σε μια κοινή δήλωση που δημιουργεί αυτό το διαθεσμικό πάνελ για τον Γαλιλαίο, Σαφώ λέει πω το Ευρωκοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Κομισιόν αναγνωρίζουν την ανάγκη συνεργασία των τριών θεσμών. Και πάλι πιστεύω πως αν το Κοινοβούλιο είναι παρόν στο, συμβου... Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί από πρώτο χέρι να βλέπει τι συμβαίνει για τα θέματα ασφάλεια, καθώς επίσης και σε σχέση με την ε, θέση σε εμπορία των διαφόρων εφαρμογών του συστήματος. Τώρα, τι θα συμβεί μετά το 2013. Ο κύριος Ρούμπιχ το ανέφερε αυτό, αλλά νομίζω είναι εξίσου σημαντικό να πούμε ότι του χρόνου ο κανονισμός απαιτεί να κάνουμε μια ενδιάμεση έκθεση, ε, αποτίμηση και να τη συνοδεύσουμε με προτάσεις για τις, τα επόμενα στάδια. Και αυτό θα το κάνουμε. Έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία ανάλυσης των επιλογών ποια θα πρέπει να είναι η διακυβέρνηση μετά από το 2013 και θα έρθει αυτό του χρόνου στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Για να δούμε δηλαδή ποια θα είναι η κατάσταση μετά το 2013 και ποιος θα είναι ο ρόλος της Κομισιόν σε εκείνη τη φάση. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία γιατί ο Πρόεδρος είπε ότι ήθελε να έχει γίνει μια πιο μακροσκελή συζήτηση για τον Γαλιλαίο. Σίγουρα το μετά το 2013 εξαρτάται από την φάση ανάπτυξη του συστήματος και των υπηρεσιών. Και αυτό είναι κάτι που θα μπορούμε να σας πούμε περισσότερα στο τέλος του χρόνου ή στις αρχές του επόμενου χρόνου όταν θα προχωρήσει ομοιοδοτικό διαγωνισμό και θα ξέρουμε ποιο ανέλαβε ποιο κομμάτι του συστήματος. Γνωρίζουμε τότε την ακριβή χρονολογία της ανάπτυξης των υπηρεσιών, την κατάσταση του προπολογισμού και θα μπορούμε να σας πούμε και περισσότερα πράγματα για την κατάσταση μετά το 2013. Επανερχόμεθα λοιπόν στα κύρια σημεία Γι' αυτό λοιπόν ζητήσαμε μεγαλύτερη ισχύ στο Διοικητικό Συμβούλιο του GSA. Θεωρούμε πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης έχει να παίξει σημαντικό ρόλο και γι' αυτό και νομίζουμε πως το καθεστώς παρατηρητή θα πρέπει να δοθεί στο Κοινοβούλιο. Επ' αυτού θα πρέπει να σας πω ήδη και θα γνωρίζετε πως το Συμβούλιο δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό στην πρόταση αυτή, στη συζήτηση μέχρι στιγμής. Και βεβαίως σε σχέση με τη διαπίστευση θα πρέπει, θέλουμε να έχουμε ανεξαρτησία στη λήψη αποφάσεων και γι' αυτό και έχουμε προτείνει αυτό τον τρόπο εργασίας για τη διαπίστευση το, της, των συστημάτων ασφάλισης. Αλλά γι' αυτό είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές ε, για τις λεπτομέρειες, για το πώς θα λειτουργήσει το σύστημα και ποια είναι η άποψη του Συμβουλίου. Θα ήταν το ιδανικό να έχουμε μια συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση από αυτού, ώστε να δούμε πώς θα στηθεί όλη αυτή η διαδικασία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πολύ κύριε Τασνόφσκι. Όχι, δεν χρειάζεται. Καλά. Ας έρθουμε στο χρονοδιάγραμμα. Προτάσεις 10 Νοεμβρίου η επόμενη ανταλλαγή απόψεων. Σχέδιο 2 Δεκεμβρίου. Τροπολογίες 9 Δεκεμβρίου. 27-28 Ιανουαρίου τροπολογίες και 4 Φεβρουαρίου τελική έγκριση στην Επιτροπή. Θα δεχθώ και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διαθέσουμε χρόνο να επανεξετάσουμε με συμμετοχή όλων των συναδέλφων που συνεργάζονται είναι κρίμα σε, μια τέτοια, σε ένα τέτοιο σημαντικό θέμα είναι παρόν μόνο εισηγητής. Να εξετάσουμε δηλαδή και τα διάφορα της κατανομής. Νομίζω ότι πρέπει να ε, είναι ενήμερη η Επιτροπή. Ας σημειώσουμε λοιπόν, κύριε Γραμματεύ, να βάλουμε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη, είτε μόνο του στις αρχές του επόμενου χρόνου, είτε μαζί με την, ε, από κοινό δηλαδή με την έκθεση κ. Καλώς λοιπόν. Στα διάφορα δεν έχω τίποτα. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλες και όλους. Και σε λίγα λεπτά, εάν συμφωνείτε, θα συνεχίσουμε με τους συντονιστάς. Και όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα.